Mes συνάδελφοι, ξεκινά η συνεδρίαση και σας υπενθυμίζω όσο φτάνουν οι τελευταίοι καθυστερημένοι καθώς και ο Γενικός Διευθυντής της ε, ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Προπολογισμό έρχεται και τον χαιρετίζω. Έχουμε μια βεβαρημένη μερίσια διάταξη και θα ξεκινήσουμε με τις σημαντικές ψηφοφορίες ιδίως σχετικά με το ε, ψήφισμα για τον προϋπολογισμό, όχι μόνον νόμος. παρακαλώ ότι όσοι μιλούν χωρίς να συμμετέχουν στη συζήτηση μπορούν να συνδιαλέγονται εκτός εθούσης. Αλλά πρώτα να πούμε χρόνια πολλά στη Γιούτα Χάου που έχει τα γενέθλιά της. Η Γιούτα έγινε 40 ετών την Παρασκευή, την περασμένη Παρασκευή. Και ε, με μεγάλη χαρά μαζί με όσους την αγαπούν ότι θέλουμε να εορτάσουμε αυτό το σημαντικό γεγονός. Καταρχήν λοιπόν τώρα για τα δικά μας η έγκριση της ημερήσιας διάταξης. για την ημερήσια διάταξη ακριβώς πριν την ε, την συνεδρίασή μας η κυρία Βέρτμαν μου απίφθινε μία παράκληση. Κυρία Βέρτμαν, μου ζητήσατε να αναβληθεί η ψηφοφορία της εκθέσεώς σας για να σας επιτρέψει να ξαναέρθετε σε επαφή με τις πολιτικές ομάδες για να δείτε αν διατηρούνται ορισμένες ορπολογίες ή όχι. Αυτό δεν είναι. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο πάλι. Σχετικά με την οδηγία της φορολογίας της ενέργειας σας το ζήτησα γιατί ε, στην πρώτη τροπολογία την οποία αναπέσυρα εκ των υστέρων λόγω της θέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διαπιστώνω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μία νέα κίνηση και προσπαθούμε να βρούμε μία συμβιβαστική λύση την οποία συζητήσαμε με τον συνάδελφο του ΕΛΚ και των σοσιαλιστών άρα παρακαλώ να αναβληθεί αυτή η ψηφοφορία για την επόμενη συνεδρίαση για να καθίσουν όλοι οι εκπρόσωποι των πολιτικών ομάδων μαζί και να μπορέσουν να καταλήξουν σε μια ενιαία διατύπωση. Ωραία. Οπότε από πλευράς προθεσμιών αυτό είναι δυνατόν και αν μπορούμε να διευκολύνουμε την επίτευξη μιας πολιτικής συμφωνίας θα αναγράψουμε αυτό το θέμα στην ημερήσια διάταξη επόμενης συνεδρίασης. Τώρα, δεύτερο θέμα που είναι η έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης της 22ης Σεπτεμβρίου που θα θεωρηθεί εγκριθήσα εάν δεν υπάρξουν παρατηρήσεις μέχρι το τέλο της ε, ε, συνεδριάσεως μετά οι ανακοινώσεις του Προέδρου υπάρχουν στο, κόκο, στο ε, Κόμπι και ξεκινάμε τις ψηφοφορίες ελπίζω ότι όλοι έχετε τις κάρτες σας ψηφοφορίας και συγχρόνως ο καθένας εκτός της κάρτας του θα πρέπει να έχει μπροστά του το σχέδιο ψηφίσματος το οποίο παρουσίασαν οι δύο εισηγητές μας η Φραντσέσκα Μπαλτσάνη και Χωσέ Μανουέλ Φερνάντες το έχω και εγώ κάπου μπροστά μου εδώ το έχετε όλοι έχετε ε, τους ε, καταλόγους της ψηφοφορίας Ο συντονιστής του ΕΛΚ δεν έχει κάρτα. Θα ε, ψηφίζει γραπτός. Βλέπετε όταν περνάτε όλοι σας την ημέρα στο διαδίκτυο δεν μας παρακολουθείτε πλέον. Πρώτη τροπολογία Μιγγέλ Πόρτας, ο εισηγητής είναι κατά ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ε, τροπολογία 2, Τζοβάνι Λαβίο, εισηγητής είναι υπέρ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ο εισηγητής είναι εδώ. Με συγχωρείτε. Φραντσέσκα, με συγχωρείς, ήρθε πολύ μακριά μου, γι' αυτό δεν σε βλέπω πια. Τροπολογία 3. Μιγγέλ Πόρτας, καταπίπτη μάλλον με συγχωρείτε, το δεύτερο μέρος της τροπολογίας. Πρώτα ας ψηφίσουμε την τροπολογία 3. Ποιος είναι υπέρ, ο την κατά. Απορρίπτεται. Άρα τίποτα δεν καταπίπτει. Η τροπολογία 4 του κυρίου Αλβάρο και άλλων υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το 5 του Μιγγέλ Πόρτα, ο εισηγητή είναι κατά. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχέ, απορρίπτεται. 6 τη κυρία Βέρτμαν, ο εισηγητή είναι κατά. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχέ, απορρίπτεται. 7. Λαβία. Ο εισηγητή είναι υπέρ. Κατά. Αποχέ, εγκρίνεται. 8 του κυρίου Πόρτα. Αντίθετο εισηγητή. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 9. Γκέραν Φέρμ, ο εισηγητής είναι υπέρ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 10. Του κυρίου Βίλμοτ. Ε, κυρίας, με συγχωρείτε. Κυρίας Βίλμοτ. Ο εισηγητής είναι κατά. Ο εισηγητής είναι κατά. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Οπότε, χες απορρίπτεται. 11 Κλαούντιο Μοργκάντι. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 12 Τζοβάνι Λαβία. Ο εισηγητής είναι θετικός. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 13 Μιγγέλ Πόρτας. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 14 από υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 15 του κυρίου Αλβάρο και άλλων ε, ε, φιλελευθέρων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 16 του κυρίου Πόρτας ο εισηγητής είναι κατά υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 17 Γκέραν Φέρμ ο εισηγητής είναι υπέρ Ποιο είναι υπέρ κατά αποχές υπάρχει μία θετική πλειοψηφία, άρα το πρώτο μέρος τροπολογίας 19 α, καταπίπτει, αλλά πρώτα ψηφίζουμε τη 18 που είναι συμβατή υπέρ κατά αποχές, απορρίπτεται. Δεύτερο μέρος της τροπολογίας 19, ο εισηγητής είναι θετικός, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 20. Μιγγέλ Πόρτας, ο εισηγητής είναι αντίθετος, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 21. Γκόραν Φέρμ, ο εισηγητής είναι θετικός, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 22. Μιγγέλ Πόρτας, που είναι συμβατό. Ο εισηγητής είναι αντίθετος, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 23 της Έλγα Τρίπελ. Ε, χωρίζεται σε τρία μέρη. Πρώτο μέρος. Μόνο οι λέξεις δίπλη. Δεν αρέσει στον εισηγητή όμως. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ευχαριστώ. Απορρίπτεται το ντύπλι και ξανα... συνεχίζουμε ε, πιο επιφανειακά. Δεύτερον, regress for energy research. Ο εισηγητής είναι υπέρ. υπέρ. Κατά. Για να κάνουμε έναν ηλεκτρονικό έλεγχο. Έχω δικαίωμα να ψηφίσω. και θα προσθέσουμε μία αρνητική ψήφο. Ανοίγει, ξεκινά η ψηφοφορία. Δεκατέσσερις υπέρ, 25, 26 κατά, απερίφθη. Και το τρίτο μέρος, έχει κάποιο νόημα το τρίτο μέρος. Έχει νόημα. Αν δεν έχουμε το πρώτο και το δεύτερο μέρος, εφόσον δεν υπάρχει τίποτα άλλο, πώς θα πούμε ε, is there for, αφού δεν ε, υπάρχει τίποτα πριν από αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, το τρίτο μέρος μπορεί να ψηφιστεί χωρίς το for, εφόσον απερίφθη ο λόγος για τον οποίο θα γινόταν αυτό. Υπέρ. η Χέλγα, πράσινη, κατά. η υπόλοιποι καταρρύπτεται επίσης, οπότε δεν έχουμε τίποτα πλέον από την τροπολογία 23. Δηλαδή, α, τρεις πύραυλοι διαφορετικοί τέστρεψαν τα τρία τμήματα της τροπολογίας. Τροπολογία 24 έλγια τρίπελ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 25. Προφορική τροπολογία του εισηγητή. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Λογικό. Αποχές. Ευχαριστώ υπάρχει μία αποχή και ε, πλειοψηφία υπέρ αυτής της τροπολογίας. Η 26 του Γκέραν αποσύρεται, 27 του Πόρτας ε, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 28 Τζοβάνι Λαβία, ο εισηγητής είναι θετικός, υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 29 του Μιγγέλ Πόρτας, αντίθετος εισηγητής, υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Το τριέντα της Αγγέλικα Βέρτμαν, ο εισηγητής είναι αντίθετος, υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. Υπάρχει μία συμβιβασική τροπολογία με α κεφαλαίο, αλλά κατόπιν του ΕΛΚ υπάρχει μία αίτηση για να ψηφιστεί χωριστά. Καταρχήν, the size reduction of youth unemployment, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος, calls nevertheless on the commission μέχρι this program. Ο εισηγητής είναι θετικός, υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. ο Σαλβατόρ μπορεί να ψηφίσει και άρα αν ε, υπάρχει πλεονάζον ΕΛΚ θα είμαι εγώ, αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει. Λίγη ψηφοφορία. 14 υπέρ, 26 κατά, απερίφθη. Τρίτο μέρος. όλσο προπόζες μέχρι εράσμους μούντους πρόγραμμα. Ο εισηγητής είναι θετικός. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Οπότε στη συμβιβαστική α, το δεύτερο μέρος απερίφθη, το υπόλοιπο ισχύει. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να θεωρήσουμε ότι οι επόμενες τροπολογίες έχουν καλυφθεί, η 31 καλύπτεται, το 32, το 33 του Γκέραν Φέρμ και του 34 της κυρίας Βέρτμαν. Ερχόμαστε τώρα στην τροπολογία 35 των φιλελευθέρων. Ο εισηγητής είναι αντίθετος, υπέρ. κατά αποχές απορρίπτεται 36 των ιδίων υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται οπότε ψηφίζουμε το 37 και αντιθέτως με ό,τι λέγεται ο εισηγητής ε, δεν σκοπεύει να το ε, ε, ενσωματώσει σαν προσθήκη. Άρα η 37 ως έχει. Υπέρ, κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Ανοίγουμε λοιπόν πάλι την ψηφοφορία 37 η οποία δεν είναι πλέον προσθήκη. Ψηφίσατε όλοι. Λίγοι. 22 υπέρ, 17 κατά, εγκρίνεται. Εγκρίθηκε το 37, το 38 καταπίπτει, που ήταν συμβατό με την 36 αλλά όχι με την 37. Αλλά ψηφίνουμε την 39 του Μιγγέλ Πόρτα, ο συγητής είναι αντίθετος. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 40 του ιδίου, υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 14 του ιδίου υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 15 του... Με συγχωρείτε, γιατί γυρίστε προς τα πίσω. Με συγχωρείτε λέει ο πρόεδρος, έκανα λάθος. Ο πρόεδρος είναι στα σύννεφα. Με συγχωρείτε και επανέρχομαι. Σελίδα 4, τροπολογία 41 του Γκέραν Φέρμ. Ο εισηγητής είναι υπέρ, υπέρ, κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 42 καλύπτεται, 43 των φιλελευθέρων υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 44 καλύπτεται του Μιγγέλ Πόρτα στο 45 της Helga Triple σε δύο τμήματα πρώτο ο τμήμα Call Zone μέχρι This Challenge ο εισηγητής είναι θετικός υπέρ κατά αποχές Νομίζω ότι οι περισσότεροι είναι θετικοί, αλλά θα κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο και εγώ δεν μπορώ πλέον να ψηφίσω, άρα δεν θα ψηφίσω. Ψηφίστε όμως εσείς και γρήγορα. Λίγη ψηφοφορία, 14 υπέρ, 26 κατά. Το πρώτο τμήμα απορρίπτεται. Υπάρχει νόημα να ψηφίσουμε το δεύτερο μέρος. Μάλιστα, λέει όχι. Οπότε, Έλγα Τρίπελ και πάλι ε, υπάρχει υπάρχουν ε, ε, πύραυλοι οι οποίοι κατέληψαν την κυρία Τρίπελ. 46 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 47 Χέλγα Τρούπελ. Ο εισηγητής είναι θετικός, υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 47 της Χέλγα. Δεν ψηφίζω, ξεκίνησε η ψηφοφορία γρήγορα και αποτελεσματικά. Λήξαμε. 19 υπέρ, 21 κατά, απορρίπτεται. 48. Γκέραν Φέρμου, εισηγητή είναι θετικό. υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και το 49. Έχουμε τώρα ε, μια συμβιβαστική β' της Φραντσέσκα, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Άρα οι δύο επόμενες ε, τροπολογίες καταπίπτουν και φτάνουμε στην 52 της Utah Haug σε δύο τμήματα. Πρώτο μέρος provides for μέχρι environmental legislation, η συγκίτρια είναι είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, and request μέχρι in a consistent way. Επίσης ο εισηγητής θετικός υπέρ. Κατά. Το δεύτερο μέρος κατά καταπίπτει. Για την 53 αντιλαμβάνουμε ότι υπάρχει μία συμβιβαστική 2α ε, στην παράγραφο 32 την οποία υποβάλλω προς ψηφοφορία. Έχετε όλοι το σχετικό έγγραφο. Είναι μία προσθήκη στην ε, ε, παράγραφο 32. Φραντσέσκα, σχολιάστε παρακαλώ. Νομίζω ψηφίσαμε στην 53. το 53. Ναι, είναι μια σωστή εντύπωση, ε, διότι αν το ερμηνεύω σωστά και διεθώστε με κάνω λάθος, προτιμώ να ψηφίσουμε τη συμβαστική σας πρώτα, αυτή είναι η στιγμή του, και αν περάσει οι τροπολογίες 54 και 57 θα καλυφθούν και 53 και 55 θα καταπέσουν. Ναι. Είναι στην ίδια, αφορούν την ίδια παράγραφο. Σύμφωνα την παράδοσή μας ψηφίζουμε λοιπόν πρώτα την πρόταση του συγητού. Αν εγκριθεί τα υπόλοιπα α, καταπίπτουν. Ξεκινάμε λοιπόν από τη συμβιβαστική β, α της υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τώρα, όλες οι άλλες α, τροπολογίες, η 53, η 54, ή 55 και 57 και 57 καλύπτονται. Όχι 56. Με την επιφύλαξη αυτού που θα μας πει ο Τζοβάνι. Πιστεύουμε εμείς ότι η τροπολογία 55 δεν καλύπτεται από το συμβιβασμό, άρα χρειάζεται να την ψηφίσουμε. 55 της κυρίας Χολμάιερ. Σύμφωνα. Όχι 57. 55. Καλώς. Συμφωνεί η συγγήτρια, είναι κατά αυτής της τροπολογίας, αλλά την ψηφίζουμε. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Χρειάζεται ηλεκτρονικός έλεγχος. Είναι μικρή η διαφορά, εγώ δεν ψηφίζω, εσείς ψηφίζετε πάντα. Ωραία. Πέρας ψηφοφορίας. 21 ψήφοι υπέρ, 20 ψήφοι κατά. Πράγματι. Η 55 εγκρίνεται και προστίθεται συμβαστική, διότι είναι συμβατή. Ψηφίζουμε την 56. 56 Helga Triple. Η συγγήτρια είναι κατά υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 57 καλύπτεται. Η 58 η 57 καλύπτεται. 58 θα πρέπει να την ψηφίσουμε. Άρα ξαναδιαβάζοντάς τη δεν ικανοποιείται η συγκήτρια, οπότε είναι κατά η συγκήτρια. δεν συνδέεται με την ε, πρώτερη ψηφοφορία. Ε, ε, υπερβάλλω τέλος πάντων. Ποιος είναι υπέρ της 58. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 58. Λοιπόν, έναρξη ψηφοφορία, εγώ δεν ψηφίζω. Πέρας. Αυτή τη φορά είναι το αντίστροφο. 20 υπέρ, 21 κατά. Η 58 λοιπόν απορρίπτεται. 59 Μιγγέλ Πόρτα, συγκίτρια είναι κατά. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 60 του κυρίου Αλβάρο, η συγκίτρια είναι υπέρ, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 61 του κυρίου Σιμάνσκι, η συγκίτρια είναι κατά, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Απορρίπτεται. 62 Μιγγέλ πόρτα, Εισηγείται είναι κατά. Υπέρ. Κατά. απόχέ, Απορρίπτεται. 63 τη κυρία Βέρτμαν. Εισηγείται είναι κατά. Υπέρ. Κατά. αποχέ, Απορρίπτεται. 64 Μιγγέλ πόρτα, Εισηγείται είναι υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 65 Γιούτα Η Εισηγείται είναι υπέρ. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Φάνουμε στη συμβαστική C της Φραντσέσκα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Οι δύο επόμενες καταπίπτουν. 68 Τζοβάνι Λαβία, εισηγήτρια είναι εναντίον. Ποιος είναι υπέρ. Κατά Αποχές απορρίπτεται το έλκυνα απομονωμένο σε αυτή την τροπολογία. 69 του ιδίου προφορική τροπολογία Β υπενθυμίζει ότι οι αυξανόμενες ανάγκε όσον αφορά τη συνεργασία με την Ασία και τη Λατινική πρέπει να γίνει να αποδεκτή στον προβλησμό 2012. Υπέρ. Κατά. Αποχές. εγκρίνεται. 70 φιλελεύθερων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Γυρνάμε τη σελίδα, σωστά αυτή τη φορά, 71 Μιγγέλ Πόρτα, η είναι κατά, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 72 Γιούτα Χάουγκ, με προφορική τροπολογία σε υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 73 του κυρίου Βαντάλεν, η είναι κατά, υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 74 Μιγγέλ Πόρτα σε είναι κατά υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 75 Γιούτα Χάουγκ προφορική τροπολογία D λατινικό που συμπληρώνει την 75 υπέρ κατά θα πρέπει να γίνει ηλεκτρονικός έλεγχος. Α, υπερθερμάνθηκε το μηχάνημα. Περιμένουμε λίγο. Λειτουργεί. Λοιπόν, έναρξη ψηφοφορία. Ψηφίστε. Εγώ δεν ψηφίζω. Πολύ του ΕΛΚ. Α. Πέρας ψηφοφορίας. 19 υπέρ, 22 ψήφοι κατά. Η προφορική τροπολογία απορρίπτεται. Συγχαρητήρια λοιπόν στη Φραντσέσκα. Ψηφίσαμε το τμήμα του ψηφίσματος που αντιστοιχούσε στην έκθεσή της. Στον ίδιο πινάκα ψηφοφοριών συνεχίζουμε. Στα άλλα τμήματα, other sections. βρίσκει τα κείμενα των συμβαστικών προτάσεων η γραμματεία. Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, 76. Μιγγέλ Πόρτας, εισηγεί τι είναι κατά, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 77. Εκεί έχουμε πρόταση κοινή του εισηγητού και του Μιγγέλ Πόρτας, ενωμένο πορτογαλικό μέτωπο, για να διαγραφεί παράγραφος 56. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 79 του εισηγητού υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 80 του κυρίου Αλβάρο που αποτελεί προστίκη αλλά καταπίπτει. Καταπίπτει. Εξαφανίζεται η προσθήκη. 81 λοιπόν. Μιγγέλ Πόρτας. Η συγκητή είναι κατά, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 82 του συγκητού υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 83 είναι συμβατή, ο εισηγητής είναι κατά, υπέρ κατά άποχες απορρίπτεται 84 Μιγγέλ Πόρτας εισηγητής είναι κατά υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 85 του ιδίου ο εισηγητής είναι κατά υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 86 είναι προφορική τροπολογία τεχνικής φύσεως του εισηγητή υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος διότι αυτή η τεχνική προφορική τροπολογία διχάζει ηλεκτρονικός έλεγχος άρχεται υπάρχει ένα μέλος του ΕΛΚ παραπάνω εκτός από μένα και άλλος ένας εντάξει Τέλος. Έληξη ψηφοφορία. 37 υπέρ, τρει ψήφοι κατά. Δεν κατάλαβα τίποτα την ταινία που είδαμε, τόσο πάνω. Λοιπόν, η 88 μετά από μάχη εγκρίθηκε. Πάλι πορτογαλική τροπολογία έχουμε του εισηγητή περ κατά τι κάνουν σοσιαλιστές εκεί πέρα 89 τροπολογία 89 Ψηφίσαμε την 88. Α, ήταν η άλλη τεχνική τροπολογία. Μάλιστα, υπάρχουν πολλές τροπολογίες τεχνικής φύσης. Λοιπόν, πρέπει να ψηφίσουμε την 88. 88 του εισηγητού. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πάμε ξανά στην 89 και την 90. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 91 του εισηγητού υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος électronique. Tous les PPE e Le vote est clos. Έλεξη ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. 24 υπέρ, 17 κατά. Εγκρίνεται. 92 Μιγγέλ Πόρτα, ο εισηγητή είναι υπέρ. Υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. 93 ο εισηγητή θέλει προφορική τροπολογία. Έχει διανεμηθεί. Είσαστε υπέρ λοιπόν της τροπολογίας αυτής. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 94. Πάλι προφορική τροπολογία τεχνικής φύσεως. 94 του συγγητή υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 95 κατά πίπτη, 96 και 97 του συγγητή υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Οι σοσιαλιστές είναι μόνοι τους στην αντίθεσή τους. Λοιπόν, οπότε καταπίπτει 98. 99 και 100 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. 101 Μιγγέλ Πόρτας. Ο είναι κατά. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Πρέπει να ψηφίσουν το 102 του εισηγητού. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 103. Αποσύρεται. 104. Με προφορική τροπολογία του εισηγητού που την έχετε γραπτός. Και μου λένε ότι έχουν ζητήσει σοσιαλιστές ξεχωριστή ψηφοφορία κατά τμήματα για την 104 το πρώτο τμήμα καλωσορίζει welcomes μέχρι mutual confidence. Για την 104. Πρώτο τμήμα. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Πρώτο τμήμα εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Από το considers θα το θεωρεί. Since then. Μέχρι το έκτοτε. Είναι υπέρ ο εισηγητής. Υπέρ υπέρ του δεύτερου τμήματος. Κατά άποχες δεν είναι ξεκάθαρο. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίζουμε, μας λείπουν ψηφοφόροι και άλλοι και άλλοι και άλλοι λείπουν. Λοιπόν, Τέλος. 21 ψήφοι υπέρ, 15 κατά, υιοθετείται και το δεύτερο τμήμα. Τροπολογία 105 του εισηγητού, ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται, μικρή διαφορά. Τροπολογία 106. Προφορική τροπολογία με προφορική τροπολογία και μία ψηφοφορία κατά τμήματα δεν καλύπτεται από την προηγούμενη αυτή η τροπολογία. Δεν υπάρχει ξεχωριστή ψηφοφορία. Δεν βλέπω split. Λοιπόν ψηφίζουμε την 106 που είναι συμβατή με την προηγούμενη. Ο εισηγητής είναι κατά. Α, είναι υπέρ, λέει ο πρόεδρος. Α, συγγνώμη. Καλεί το Προεδρείο να μην συνδέσει τις αμοιβέ των μελών με τον πληθωρισμό. Φιλανδική τροπολογία, περίφημη. Αυτή είναι η προφορική τροπολογία. Με αυτή την τροπολογία λοιπόν, ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 106. Πάμε στην 107. Καλύπτεται. 108. Δεν καλύπτεται η 108. Ο εισηγητής είναι κατά. Υπέρ. Α, συγγνώμη, λέει ο πρόεδρος. Εκατόν Πρώτο τμήμα. Urges μέχρι elections. Καλύπτεται αυτό. Δεν ξέρουμε. Ψηφίζουμε λοιπόν. Γιατί δεν ξέρουμε αν καλύπτεται. Λοιπόν, για το πρώτο τμήμα του εισηγητή που είναι κατά. Ποιο είναι υπέρ για το πρώτο τμήμα. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος, δεν είναι ξεκάθαρο. Πρώτο τμήμα τη 108. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι υπέροχα. Αποτέλεσμα. 18 υπέρ, 21 ψήφοι κατά. Απορρίπτεται το πρώτο τμήμα. Το δεύτερο τμήμα έχει νόημα. To ensure μέχρι allowance. Έχει νόημα. Ο εισηγητής είναι κατά. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται επίσης δεν υπάρχει τίποτα πια από την 108, έχει μείνει. 109 της κυρίας Βίλμοντ. Το εισηγητής είναι κατά, υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. 110 του εισηγητού, προφορική τροπολογία. Ναι. Καλύπτεται. Εξαφανίζεται 110, 111. Η 107 είχε εγκριθεί, άρα καταπίπτει 111. Δεν φτάσαμε κάνω λάθος. 112 και 113 υπάρχει συμφωνία του εισηγητού με τους σοσιαλιστές που είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 114 αποσύρεται. 115 Γκόραν Φέρμ, ο εισηγητής είναι κατά. Καλύπτεται λέει ο πρόεδρος. Καλύπτεται. 116 δεν καλύπτεται. Με προφορική τροπολογία του συγγητού να διαγράψουμε τον παιδικό στα accounting Office υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 117 του συγγητού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 118 Γκέραν firm είναι κατά εισηγητής που είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 119. Γκέραν Φέρ με προφορική τροπολογία του φυγητού. Ο είναι υπέρ. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 120. Των φιλελευθέρων που είναι συμβατή με προφορική τροπολογία του συγητού. Ποιος είναι υπέρ. Κατά 120. Καταπίπτει 120 λόγω της 119. Καλώς. 121. Καταπίπτει επίσης. Χολμαϊρ. Καταπίπτει. Καταπίπτει. 122. Γκέραν Φέρμ. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 123 του εισηγητού και, της κυρίας, και του κυρίου Μουργκάντη. Υπέρ, κατά, ηλεκτρονικός έλεγχος. 123, ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίζουμε, ψηφίζουμε, πέρας, ψήφισαν όλοι. Αποτελέσματα 22 υπέρ 17 κατά εγκρίνεται οπότε 125 καταπίπτει. Ψηφίζουμε την 126 Γκόραν Φέρμ, ο εισηγητή είναι υπέρ. Υπέρ, κατά, Αποχέ εγκρίνεται. 127 υπέρ, κατά, Αποχέ εγκρίνεται. 128 υπέρ, κατά, Αποχέ εγκρίνεται. 129 Μπορούμε να ψηφίσουμε 129, 130, 131 μαζί του εισηγητού υπέρ υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται και τρεις 132 Helga εσύ γιατί είναι υπέρ, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 133 αποσύρθηκε 134 με προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται οπότε οι, επόμενες, οι δύο επόμενες καταπίπτουν πάμε στην 137 Γκουαλτιέρη και Βον με δύο, σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα σταματά στην κυρία Άστον και ικανοποιεί τον εισηγητή. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, από το therefore μέχρι lifted, ο εισηγητής είναι κατά, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, πρέπει να γίνει ηλεκτρονικός έλεγχος, για το δεύτερο τμήμα της 137, έναρξη ψηφοφορίας ηλεκτρονικού ελέγχου. Πέρας. Τέλος ψηφοφορίας. Τι λέει, ποιο είναι το αποτέλεσμα. 16 υπέρ, 25 κατά, το δεύτερο τμήμα απορρίπτεται. 138 του κ. Φερνάντες υπέρ, κατά, ηλεκτρονικός έλεγχος. Λυπούμε για την 138 και εδώ ηλεκτρονικός έλεγχος. Ξεκινάμε. Πέρας ψηφοφορίας. 23 υπέρ, 16 κατά, εγκρίνεται. 139 που είναι συμβατή με την 138 εισηγητής είναι υπέρ, υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται 140 του εισηγητού υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 141 δύο τμήματα έχουμε πρώτο τμήμα remarks μέχρι commission ο εισηγητής είναι υπέρ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα therefore μέχρι reinstated ο εισηγητής είναι κατά υπέρ ηλεκτρονικός έλεγχος δεύτερο τμήμα της 141 ψηφίστε Έληξη ψηφοφορία. 16 υπέρ, 24 ψήφοι κατά, απορρίπτεται. 142 του ηγητού είναι υπέρ. Λοιπόν, υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται 143 ο συγητής. Α, καταπίπτει. Πριν την τελική ψηφοφορία. Ήθελα να υπενθυμίσω ότι το περιεχόμενο των γνωμοδοτήσεων που εκδίδονται από τις ΑΦΚΟ, ΑΦΕΤ, ΑΓΚΡΙ, ΕΚΟΝ, Απασχόλησης, ΕΜΒΙΜΚΟ, ΙΝΤΑ, ΙΤΡΕ, ΛΥΜΠΕ, ΠΕΣ, ΠΕΤΗ, ΡΕΖΙ, ΤΡΑΝΣ έχουν ληφθεί υπόψη στο βαθμό του δυνατού, όσο το δυνατόν περισσότερο, από το σχέδιο της εκθέσεως, του συμβιβασμούς και της ψηφοφορίας λαμβάνοντας υπόψη τη διαβούλευση που έλαβε χώρα μεταξύ εισηγητού με τους δικευμένους εισηγητές αυτών των επιτροπών. Άρα το περιεχόμενο θεωρείται ότι καλύπτει ψηφοφορία της Επιτροπής Προϋπολογισμών και θα προσαρτηθεί στο ψήφισμά μας. Τελική ψηφοφορία όσον αφορά το ψήφισμα αυτό θα γίνει ηλεκτρονική ψηφοφορία αλλά δεν μπορώ να ψηφίσω. Θα ήθελα να ψηφίσω. Να δω αν περισσεύω. Α, δεν περισσεύω. Μπορώ να ψηφίσω. Θα ψηφίσω. Ψήφισα. Σταματάμε την ψηφοφορία. Αποτελέσματα. 34 ψήφοι υπέρ, 7 κατά, καμία αποχή. Μπράβο. Συγχαρητήρια κυρία και κύριε εισηγητά. τώρα σας προτείνω να περάσουμε στο σημείο 9 που θα είναι πολύ γρήγορο. Πρόκειται για την έκθεση Μπέγκε για την κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας υπέρ της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας και του προγράμματος πλαίσιο για την έρευνα. Μία ψήφος. Μία ψηφοφορία. Αγαπητοί συνάδελφοι, ηρεμήστε λίγο. Πρόκειται για μια έκθεση την οποία χρειαζόμαστε μαζί με τις ψηφοφορίες για τον προπολογισμό, γιατί θέλουμε να ξεκινήσει η διαδικασία κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας, ώστε να χρηματοδοτηθούν τα πλεονάσματα πιστώσεων που χρειαζόμαστε σε δύο κατηγορίες, την 1α και την 4 πρέπει να κινητοποιηθεί το μέσο ευελιξίας. Για να γίνει αυτό, αυτό σημαίνει αναθεώρηση των δημοσιονομικών προοπτικών, Όχι, διορθώνει ο πρόεδρο. Αυτό σημαίνει την προσφυγή στη διάταξη της Διοργανικής Συμφωνίας που προβλέπει την κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας. Έχουμε ένα ειδικό εισηγητή που είναι ο Ράιμερ Μπέγγε, αλλά δεν είναι παρόν. Όμως, έχει συμφωνήσει με τη Φραντσέσκα. Και η Φραντσέσκα θα μας κάνει την έκθεση και αμέσως μετά θα ψηφίσουμε. Φραντσέσκα. Μετά από την συνεδρίαση των συντονιστών είχα μία σύντομη ε, συνομιλία με τον συνάδελφο Μπέγκε σε σχέση με τον ε, τίτλο της ε, έκθεσης και την παράγραφο 2. Και συμφωνήσαμε για την ιδέα της αλλαγής της αναφοράς στο πρόγραμμα πλαίσιο έρευνας να το ονομάσουμε Στρατηγική 2020 στον τίτλο και στο εσωτερικό της έκθεσης στην παράγραφο 2 έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια ένδειξη για το πεδίο χρήσης ε, του μέσου ευελιξίας ευρύτερο και ε, καθώς ε, η στρατηγική 2020 περιλαμβάνει το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και έτσι αν το κάνουμε αυτό αυτή την αλλαγή μπορούμε να μιλήσουμε για ένα πεδίο χρήσης ευρύτερο. Σας ευχαριστώ. Ποιοι είναι υπέρ αυτής της έκθεσης όπως τροποποιήθηκε προφορικά. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Πάντα είναι κατά. Αποχές εγκρίνεται. Να θυμίσω ότι το σχέδιο δράσης μας, η στρατηγική μας, περιλαμβάνει την ψηφοφορία στην Επιτροπή Προπολογισμού. Το έκαναμε, εγκρίναμε την έκθεση ε, του Ράιμερ, αλλά δεν θα υποβάλουμε στην Ολομέλεια την έκθεση αυτή παρά μόνο στην ε, φάση της τελικής συμφωνίας για τον προπολογισμό, δηλαδή μετά τη συνδιαλλαγή. Είναι καλύτερη μέθοδος ώστε να χρησιμοποιήσουμε καλά το όπλο των διαπραγματεύσεων ε, για το μέσο ευελιξία. Μπορούμε τώρα να επανέλθουμε στη ψηφοφορία του σχεδίου διορθωτικού προπολογισμού υπαριθμών 5 για την έκθεση της Helga Τρούπελ για τον επόπτη προστασίας δεδομένων και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Υπάρχουν δύο τροπολογίες. Η πρώτη αφορά το οργανόγραμμα, μια τροπολογία της συγχύτριας, ποιοι είναι υπέρ. κατά, αποχές, εγκρίνεται. Επιτάχουμε στο άρθρο 2, τροπολογία 1 του Ρομπέρτο Γκουαλτιέρη. Α, έχει αποσυρθεί. Έχει αποσυρθεί γιατί καλύπτεται από το νέο κείμενο. Μάλιστα, ωραία. Τελική ψήφος τώρα για την έκθεση υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πρόκειται για ένα θέμα που μπορούμε να βάλουμε στην ημερήσια διάταξη του επόμενου, επόμενου τριμερού διαλόγου με το ε, Συμβούλιο, δηλαδή στις 16 Νοεμβρίου. Πρέπει να ψηφίσουμε πρώτα στην Ολομέλεια και μετά θα το συζητήσουμε στις 16 Νοεμβρίου. Θα σας το επιβεβαιώσουμε κιόλας η έκθεση για την έκθεση Βέρτμαν αναβλήθηκε, η ψηφοφορία με συγχωρείτε. Ερχόμαστε στο σημείο 12 όπου έχουμε διάφορα ντοσιέ για το προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση. Η Μπάρμπαρα Ματέρα θα μας τα παρουσιάσει και θα τα ψηφίσουμε. Eh. Μάλιστα, Πρόεδρε. Ναι, Μπάρμπαρα. Έχουμε μία μόνο ψηφοφορία για την ε, έκθεση Ρενό, που είχαμε αναβάλει την περασμένη φορά, επί της οποίας είχαμε μια μακρά συζήτηση με την Επιτροπή για την Απασχόληση ε, σκεφτήκαμε διάφορες λύσεις, εν πάση περιπτώσει θα τα πείτε αυτά, θα δώσουμε το λόγο στην Κομισιόν και μετά βεβαίως σε όσους το επιθυμούν, γιατί δεν είχαμε πραγματική συζήτηση επί της ουσίας. Θα προσπαθήσουμε να διευκρινίσουμε κάπως τις θέσεις των διαφόρων, να δούμε τι μας συμβουλεύει η Επιτροπή Απασχόλησης, να δούμε ποια είναι η θέση της Επιτροπής και μετά θα το ψηφίσουμε. Η συγγήτρια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λοιπόν, εδώ παρεμβαίνω για αυτή την έκθεση την οποία εξετάσαμε νωρίτερα μετά από αίτημα της Επιτροπής Απασχόλησης να γίνουν κάποιοι έλεγχοι για τις διασκέψεις κορυφή, ε, για τα συμβούλια της Ρενό. Σας συνθυμίζω ότι είναι από τα πιο σημαντικά αιτήματα που έχουν γίνει για αυτό το ταμείο ε, από τότε που δημιουργήθηκε. Πρόκειται για ποσά της τάξης των 24 εκατομμυρίων ευρώ. Μια βοήθεια που θα τα πάρουν 3.500 ε, εργαζόμενοι. Το θέμα αυτό λοιπόν είναι λεπτό και έχει παρουσιαστεί από την ε, Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και από την Πρόεδρό της, την κυρία Μπερές αφορά την βήμαχη ε, κατάσταση 71 πρώην εργαζομένων της Ρενό, οι οποίοι επέλεξαν ένα πρόγραμμα πρόορης εθελοντικής σύνταξης το 2008. Αυτοί λοιπόν οι πρώην υπάλληλοι μετά από την αύξηση του έτους συνταξιοδότησης με νομοθεσία που έγινε το 2010 στη Γαλλία, από τα 60 δηλαδή στα 62, έμειναν έξω από την αγορά εργασίας. Αποκλείστηκαν και άρα δεν μπόρεσαν να συμπληρώσουν τα απαραίτητα εργάσιμα χρόνια για να μπορέσουν να συνταξιοδοτηθούν. Στην γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ζητάν, ζητούν εκεί από την Επιτροπή Προπολογισμού να βάλει σε αναμονή ένα μέρος των κονδυλίων έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορέσει να ενεργήσει με, πρώτα με έναν έλεγχο στην Ρενό, δηλαδή έναν έλεγχο, μια επαλήθευση ώστε να εξασφαλίσει ότι η εταιρεία έχει προβεί στα καλύτερα δυνατά μέτρα τόσο από νομική άποψη όσο και από οικονομική, ώστε να μπορέσει να στηρίξει του εργαζόμενου, να εγγυηθεί τα συνταξιδοτικά του δικαιώματα και τι αποζημιώσει του πάνω απ' όλα για αυτού του εργαζόμενου που επέλεξαν την εθελοντική πρόορη συνταξιοδότηση. Ανέκαθεν, η συνεργασία τη Επιτροπή Προπολογισμών με την Επιτροπή Απασχόληση και Κοινωνικών Υποθέσεων είναι σαφή. Εμεί πάντοτε συμβαδίζουμε μαζί του και εν γέννη στα τελευταία χρόνια δεν είχαμε ποτέ δυσκολίες και προβλήματα. Ε, και θα ήθελα και σε αυτή την περίπτωση να είμαστε ενωμένοι και συμπαγείς. Διότι η Επιτροπή Προπολογισμού, δηλαδή σε αυτή την περίπτωση εγώ ως εισηγήτρια για αυτό το Ταμείο για την Επιτροπή Προπολογισμού, είμαι υποχρεωμένη να θυμίσω ποια είναι τα καθήκοντά μας και οι υποχρεώσεις μας. Δηλαδή να ε, μείνουμε στον κανονισμό του Ταμείου της ε, προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση που δεν προβλέπει τέτοια ποσά που θα πρέπει να δοθούν στις κεντρικές κυβερνήσεις αλλά και στη συνέχεια στις εταιρείες που ζήτησαν την ενεργοποίηση αυτού του Ταμείου και επίσης στην ιστορία του ταμείου αυτού δεν έχει ζητηθεί έλεγχος από πλευράς κομισιών, δεν έχει ζητηθεί επαλήθευση για τη χρήση των ποσών αυτών που φτάνουν στα εταιρείε. Εγώ ανέκαθεν είπα και θύμισα ότι τα χρήματα αυτά δεν φτάνουν στις εταιρείε τις ίδιες, δεν ε, αναδιαρθρώνουν την εταιρεία, αλλά φτάνουν στους εργαζόμενους. Είναι ένα είναι ε, ταμείο το οποίο έχουμε ορίσει πολλές φορές, είναι ένα ταμείο αλληλεγγύης στην ουσία, διότι στηρίζει την επανένταξη στην αγορά εργασίας εργαζομένων οι οποίοι είχαν μείνει εκτός. Πολιτών, Ευρωπαίων πολιτών δηλαδή, που έχασαν τη δουλειά τους. Και αυτό το αίτημα ελέγχου, λοιπόν, δεν είναι δυνατόν ε, εγώ σε αυτό επιμένω και στον κανονισμό. Ξέρω όμως ότι είναι παρούσα στην αίθουσα η Επιτροπή και θα ήθελα να το ζητήσω περαιτέρω επεξηγήσεις, αν το επιτρέπετε και εσείς Πρόεδρε, σε σχέση με τα όσα μόλις είπα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω κάποιον άλλο να ζητά το λόγο. Προτείνω να δώσουμε πρώτα το λόγο στην κυρία Γκριέ. ο κύριος Νταρντέν πρώτα. Ο κύριος Νταρντέν, μετά η κυρία Γκριέ, μετά η Τρούπελ, ο κύριος Ρικέ και μετά η Επιτροπή που αντιπροσωπεύει το Γενικό Διευθυντή. Ο κύριος Νταρντέν. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Μπάρμπαρα εξήγησε την κατάσταση που είναι μια κατάσταση πρωτότυπη, δεν την έχουμε ξανασυναντήσει και είναι, λίγο εύκολο να λέει κανείς ότι επειδή δεν έχει συμβεί παλιότερα δεν μπορούμε και να το κάνουμε. Η κατάσταση είναι κάπως ιδιαίτερη και ε, σχετίζεται με την εξέλιξη της νομοθεσίας στην Γαλλία. Αφορά κάποιες δεκάδες και κάποιες μάλλον εκατοντάδες εργαζομένων και μην ξεχνάμε το βασικό μας στόχο που τον θύμισε εξάλλου η Μπάρμπαρα, δηλαδή να βοηθήσουμε τους εργαζόμενους. Έχουν γίνει διάφορες επαφές ανάμεσα στην Επιτροπή Απασχόλησης, στην επιχείρηση, τα συνδικάτα, δηλαδή τους εκπροσώπους των εργαζομένων και πιστεύω ότι αυτό που υιοθετήθηκε στην Επιτροπή Απασχόλησης θα έπρεπε να αντικατοπτριστεί εδώ στην ε, απόφαση της Επιτροπής ε, προϋπολογισμού. Γι' αυτό και με την Εστέλ καταθέσαμε αυτές τις προφορικές τροπολογίες και σας ζητούμε να ληφθεί αυτή η απόφαση που είναι ναι, που είναι πρωτότυπη και νέα, αλλά να συνδεθεί ένα τμήμα της βοήθειας με την εξέλιξη της υπόθεσης αυτής στην Ρενό. Σας ευχαριστώ. Εστέλ, θέλετε να συμπληρώσετε. Ναι. Να σας πω ότι δεν είναι απλώς λεπτό θέμα, είναι ένα θέμα εξαιρετικά σοβαρό. Ο κύριο Σταβάρα, που είναι γενικός διευθυντή τη Γαλλίας για τη Ρενό ε, είπε ότι μόνο στο εργοστάσιο της Σαντουβίλ υπήρχαν 192 άνθρωποι, 192 ε, εργαζόμενοι. Θα μπορούσα να σας το πω αν είχατε δεχτεί την, το αίτημά μα για ραντεβού. Έχουμε νούμερα εξαιρετικά διαφορετικά από αυτά που έχετε εσείς και μάλιστα νούμερα που προέρχονται από την ίδια την εταιρεία. Αυτό που μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή η δυσκολία είναι ότι οι προθεσμίες εισαγγελικέ, όπως τις γνωρίζουμε, που είναι η, αυτή που θα ωφεληθεί από επιστροφή κονδυλίων. Επιστροφή κονδυλίων, πράγμα το οποίο στην ουσία ε, κάνει τον κόσμο να αφισβητεί για το κατά πόσο αυτά τα χρήματα θα τα πάρουν οι εργαζόμενοι και γι' αυτό και υπάρχει μια σύγχυση σε εθνικό επίπεδο για τα χρήματα αυτά που θα ωφελήσουν την επιχείρηση και όχι τους εργαζόμενους σε αυτή την περίπτωση και επιπλέον αφήνει πάνω από 300 ανθρώπους στην κατάσταση που εσείς είπατε. Ε, και έχουμε και τους καταλόγους με τα ονόματα αυτών των ανθρώπων. Εγώ νομίζω ότι σε αυτή την υπόθεση θα πρέπει να έχουμε ε, πιο ευρεία άποψη. Η υιοθέτησή του γίνεται με ειδική πλειοψηφία στην Ολομέλεια και γι' αυτό και θα ήταν καλύτερο να βρούμε μια λύση εδώ στην Επιτροπή Προπολογισμού που να ταιριάζει σε όλους, να μην είναι ακραία βεβαίως, αλλά να μπορούμε να κάνουμε ένα βήμα και προς τους εργαζόμενους. Εγώ επιμένω για αυτό το θέμα. Αν δεν ληφθούν κατά κάποιο τρόπο υπόψη αυτές οι τροπολογίες που δέχομαι να το εξετάσω μαζί σας, δεν νομίζω πώς θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε και στην ε, εκχώρηση αυτών των χρημάτων. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Ρίκικε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να χωρίσουμε τα όσα μας ανησυχούν ε, σε ανθρώπινο επίπεδο και σε κοινωνικό επίπεδο από αυτά που είναι δυνατόν και ε, επιθυμητό να γίνουν. Θα πρέπει να πούμε ότι περίπου 200 εργαζόμενοι βρίσκονται σε κατάσταση που δεν είναι σύμμορφη με τα όσα προβλέπονται από αυτήν εδώ την περίπτωση λόγω της αλλαγής της ε, νομοθεσίας στη Γαλλία, αλλά να θυμίσω τα εξή. Καταρχήν, δεν έχουμε το δικαίωμα ούτε μπορούμε να, να επιβάλλουμε έλεγχο στην επιχείρηση και άρα λοιπόν αυτό το αίτημα της Επιτροπής Απασχόλησης δεν αντιστοιχεί σε καμία νομική δυνατότητα, νομικά αποδεκτή δυνατότητα έπειτα. Ο δημοσιονομικό κανονισμός απαγορεύει το να δοθεί ένα τμήμα του ποσού και όχι το άλλο, δηλαδή είναι όλα ή τίποτα. Τρίτον, έτσι όπως έχει παρουσιαστεί αυτή η υπόθεση από, από το γαλλικό κράτος λαμβάνει υπόψη τα όσα υπόθηκαν. Ότι δηλαδή ιδιαίτερα, τα ιδιαίτερα προσόντα αυτών των εργαζομόνων έχουν ε, ξεχαστεί και ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη στο πλαίσιο της επικουρικότητας από το γαλλικό κράτος. Αλλά εμείς δεν μπορούμε να υπερβούμε τον δημοσιονομικό κανονισμό, δεν μπορούμε να ε, ενεργήσουμε εμείς τη θέση του γαλλικού κράτους. Και κάτι ακόμα το οποίο άκουσα και με εντυπωσίασε είναι η απειλή ότι θα μπορούσαμε να αντιτεθούμε μέσω της ειδική πλειοψηφίας για πρώτη φορά και ενδεχομένως ε, από τους ίδιους ε, τους ε, βουλευτές της ενδιαφερόμενης χώρας στην εκχώρηση αυτών των κονδυλίων του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση που είναι όλα, όπως είπαμε, εντάξει και σύμμορφα με την νομοθεσία. Υπάρχει η υπόθεση των 200 εργαζομένων της Ρενό που θα πρέπει να ρυθμιστεί από το γαλλικό κράτος. Εμείς δεν μπορούμε παράνομα να κρατήσουμε σε ομοιρία ένα τμήμα του Ταμείου για να βαρύνουμε στην απόφαση του κράτους, του γαλλικού κράτους ή οποιοδήποτε άλλο. Σας ευχαριστώ. Το λόγο τώρα θέλει η κυρία Χέλγα Τρούπελ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Από δικιά μου άποψη θα συμφωνούσα ότι η περίπτωση αυτή είναι πολύ λεπτή και νομίζω όπως είπε και η Μπάρμπαρα Ματέρα ότι στο παρελθόν πάντοτε έχουν υπάρξει οι ίδιες ερμηνείες από την Επιτροπή Προπολογισμού και την Επιτροπή Απασχόλησης. Αυτό όμως δεν είναι δεδομένο τώρα, άρα υπάρχουν και άλλα προβλήματα όπως και άλλες παρεφερείς περιπτώσεις. Πρέπει να είμαστε λοιπόν πολύ προσεκτικοί και προφανώς χρειαζόμαστε περισσότερες διευκρινήσεις και ε, δεν επαρκεί να λέμε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα και πρέπει απλώς να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι σωστό. Ευχαριστώ. Και τελικά η Ίνγκε Χέσλερ. Ευχαριστώ. Πάντοτε είμαι ε, καχύποπτη όταν μας λένε ότι κάτι δεν επιτρέπεται από το δημοσιονομικό κανονισμό. Κάποιος θα θέλει λοιπόν να μου το εξηγήσει διότι εγώ δεν καταλαβαίνω τι μας επιτρέπει ο δημοσιονομικός κανονισμός. Ευχαριστώ. Κύριε Γενικέ Διευθυντά, μας λέτε πώς βλέπει το θέμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι κάτι παραπάνω από ένα συνέστημα. Εγώ θα σας κάνω μία ανάλυση την οποία μπορούμε να παρουσιάσουμε στην περίπτωση αυτή. Σεβόμαστε απολύτως τα διάφορα θέματα τα οποία εθίγησαν και στην πραγματικότητα ε, η νομική, η νομική πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική διότι αφενός το άρθρο 13 του κανονισμού του Ταμείου μας υποχρεώνει να πληρώσουμε εφάπαξ σε μία δόση. Δεν μπορούμε δηλαδή να σπάσουμε σε δύο ή περισσότερες ε, ε, ε, δώσει στο θέμα και επιπλέον όπως ελέγχθη δεν έχουμε καμία αρμοδιότητα για να προβούμε σε έναν οικονομικό έλεγχο για τον τρόπο με τον οποίο η επιχείρηση Ρενό προχωρά στην κατανομή των ποσών που πρέπει να αποπληρώσει. Όπως είπαμε αυτά έχουν εξεταστεί η ε, αίτηση έγινε αποδεκτή. Επεμβαίνουμε για ένα τμήμα των πόρων και εκεί περιορίζει την παρέμβαση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Το αρνητικό στοιχείο σε όλα αυτά και ε, αυτό είναι το αρνητικό στοιχείο και νομίζω ότι εδώ θα σταματήσω. Ευχαριστώ. Είναι μια υπόθεση η οποία όντως είναι περίπλοκη. Το έχω συζητήσει με την Φερμόν Σπερές, με την κυρία Γκρελιέ και εγώ προσωπικά προσπάθησα να δω εάν μπορούσαμε να διερευνήσουμε ε, μία λύση σύμφωνα με την οποία για να διευκολύνουμε την, ευκολύνουμε την ε, κατάσταση των εργαζομένων οι οποίοι είναι σε ε, δυσχερή θέση λόγω ακριβώς της παγκοσμιοποίησης αν μπορούσαμε να κινητοποιήσουμε ορισμένες πιστώσεις οι οποίες θα έμεναν σε ένα απόθεμα ή θα προβλεπόντουσαν σε δύο φάσεις και η Επιτροπή όπως και οι υπεύθυνοι μας λέγουν αυτό δεν γίνεται, δεν μπορεί ούτε να τοποθετηθεί σε απόθεμα ούτε να πληρωθεί σε δύο δόσεις. Έχει όμως υπάρξει μία με ευρεία συζήτηση από τον εκπρόσωπο της Ρενό με την υπεύθυνη της Επιτροπής Απασχόλησης και φαίνεται ότι το πρόβλημα ουσιαστικά το οποίο αντιμετωπίζουν ορισμένοι εργαζόμενοι και ο αριθμός τους διαφέρει αναλόγως του ομιλούντος ε, ε, αναφέρεται εις ε, το, το, ποσό μετά τη συμφωνία μεταξύ της Ρενό με τα συνδικάτα και την αλλαγή της γαλλικής νομοθεσίας διότι τα βοηθήματα που οι ενισχύσεις που δόθηκαν από το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης για την ανακατάταξη και για την επαγγελματική η δεν εφήγησαν από αυτές ε, τις ρυθμίσεις. Οπότε εγώ δεν βλέπω τι μπορούμε να κάνουμε, ούτε να δεχθούμε, ούτε να απορρίσουμε συλλήβδιν όπως λέει η, η Πρέπει δηλαδή εκ των δύο να διαλέξουμε το ένα και ε, διαφορετικά θα δεσμεύσουμε αυτή την ενίσχυση του Ταμείου Παγκοσμιοποίησης ε, και για να έχουμε σε άλλο επίπεδο ε, υποχωρήσεις εκ μέρους της επιχείρησης. Είναι δηλαδή ένα κάπως περίπλοκο και λεπτό θέμα. Περαιτέρω, η συγγήτρια μας παρουσίασε τη θέση της. Έχουμε τρεις ε, προφορικές τροπολογίες τις οποίες παρουσίασε ε, ο κύριος Νταρδέν και η κυρία Γκρελιέ και αναλαμβάνουμε ότι ο εισηγητής δεν συμφωνεί. Άρα αυτές οι τροπολογίες είναι ουσιαστικά προσθήκες και προσθέ, ε, προστίθενται πότε. θα τις αντιμετωπίσουμε ε, σύμφωνα με το κείμενο. Στην πρώτη παράγραφο έχουμε δύο τροπολογίες. Μία γραπτή τροπολογία της κυρίας Γκρελιέ Νταρντέν. Ε, ο εισηγητής είναι κατά, υπέρ, κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3 με την προφορική τροπολογία των ιδίων. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, πάλι τα ίδια απορρίπτεται. Τροπολογία 4 με, τον ιδίων υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5. Ρολάντα Πάξα, ο εισηγητής είναι υπέρ. Επίσης το 5, 6, 7 μπορούν να ψηφιστούν μαζί. Όχι. 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 7 εγκρίνεται. 7. Ε, Ο εισηγητής είναι υπέρ. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται επίσης. 8 της κυρίας Γκρελιέ και Φρεντερίκ Νταρντέν ε, που λέγεται ότι ε, ε, προσέβησε εργαζόμενους συμβασιούχους η απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα της ιδίας τροπολογίας, ο εισηγητής έχει την ίδια θέση υπέρ, κατά, εδώ όμως θα κάνω έναν ηλεκτρονικό έλεγχο. Πρόκειται για το δεύτερο τμήμα το οποίο ελέγχεται ηλεκτρονικά. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. 22 υπέρ 16 κατά το δεύτερο τμήμα εγκρίθηκε. Τροπολογία 9 των φιλελευθέρων. Ο εισηγητής είναι κατά. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 10. Πάξας. Ο εισηγητής είναι αντίθετος. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Επανερχόμαστε λοιπόν στην δεύτερη προφορική τροπολογία Γκρελιέ Νταρντέν για ε, τον ε, οικονομικό έλεγχο υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Τροπολογία 3 των ιδίων υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Ε, η τροπολογία 1 αλβάρο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικός έλεγχος κατευθείαν ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Λίγοι. 16 υπέρ, 20 κατά. Οπότε δεν θα γίνει έκθεση. Δεν υπάρχει δηλαδή απόφαση. Ε, τότε δεν υπάρχει μεταφορά και πληρωμή και ο καθένας θα αναλάβει τις ευθύνες του. Προχωράμε τώρα στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Πρέπει να ψηφίσουμε ε, πληρωμές, μεταφορές. Στο σημείο 13... Όχι, η συντονία έχεις πληρωμή, έχεις μεταφορά. Όσον αφορά τις μεταφορές, μας ζήτησαν να μεταφερθούν μία μεταφορά υπαριθμών 34 η αίτηση αυτή η οποία σας δώσει αναφέρθηκε εις ε, το έμβασμα το οποίο κάνει κάθε φθινόπορο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο συγητής προτείνει να ψηφιστεί στις 7 Νοεμβρίου γιατί εντωμεταξύ θα έχουμε λάβει το διορθωτικό προπολογισμό υπαριθμών 6 και ε, την ε, πρόβλεψη του προϋπολογισμού που μας ανέφερε ε, ο εισηγητής την περασμένη εβδομάδα. Θα έχουμε δηλαδή μια πιο γενική εικόνα. Συμφωνείτε κύριε Γενική Διευθυντά. Ωραία. Δεν θα ψηφίσουμε το έμβασμα 22 που αναφερόταν εις την ενίσχυση της Ρονό την οποία απορρίψαμε. Όσον αφορά όμως το 29 προτείνεται να ψηφιστεί την επόμενη εβδομάδα διότι ε, συνδυάζεται με μία άλλη κίνηση για την Αυστρία που θα μας παρουσιάσει η κυρία Ματέρα όταν τελειώσουμε τις ψηφοφορίες. Όσον αφορά την 36, ε, ζητήθηκε κατόπιν ετήσως του εισηγητή Αλφόνση ε, μία αναβολή εφόσον αναφέρεται στη Συμφωνία Αλληλείας μεταξύ Μαρόκου και Ευρωπαϊκής Ενώσεως και η ε, μεταφορά θα πρέπει να γίνει μαζί με την γνωμοδότηση, Οπότε αυτό πρόκειται να γίνει 8 Νοεμβρίου και θα ψηφίσουμε σε 7 Νοεμβρίου. Το ίδιο και με το 41 που είναι μια άλλη κινητοποίηση του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και θα ψηφιστεί μαζί με την έκθεση Ματέρα. Όσον αφορά τους προπολογισμού άλλων οργανισμών. Έχουμε δύο, ένα για τον διαμεσολαβητή και δύο δεύτερον για το ε, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και η κυρία Τρούπελ παρουσιάζει τα θέματα αυτά. Ο μεσολαβητής έχει μία γραμμή στον προϋπολογισμό που δεν έχει καλυφθεί όσο γρήγορα θα μπορούσε για να αφομοιωθεί και ζητά να υπάρξει ε, και άλλη διότι έχει διάφορες επιπλέον δαπάνες το ποσό είναι 140.000 ευρώ και ε, εγώ ε, δεν αντιτίθεμαι σε αυτή τη μεταφορά. Θέλετε πρώτα να συζητήσουμε αυτό ή να συζητήσουμε κατευθείαν και το δεύτερο. Καταρχήν για τον διαμεσολαβητή. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Ποιος είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Όσον αφορά το δικαστήριο. Το δικαστήριο θέλει να μεταφέρει 171.000 ευρώ εις τα λειτουργικά έξοδα για συμβασιούχους στο προσωπικό και 50.000 ευρώ από την πληροφόρηση στα διοικητικά έξοδα και στη σχετική γραμμή και 6.000 ευρώ για τα κτίρια. Το δικαστήριο μας έχει εξηγήσει κάθε μεταφορά και νομίζω ότι αυτά είναι πιστικά και δεν σκοπεύω να σας προτείνω να μην αντιταχθούμε σε αυτή τη μεταφορά. Ευχαριστώ. Διπλό αρνητικό σημαίνει ένα θετικό. Είμαστε, είμαι υπέρ, λέει η κυρία Τρυπέλη. Στο κλασικό γαλλικό θέατρο ήταν έτσι. Δεν σε μισώ, σημαίνει σε λατρεύω στο θέατρο. Λοιπόν, ποιο είναι υπέρ, Έλγα. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ωραία. Τελειώσαμε με τις ψηφοφορίες. Έχουμε ακόμα τρεις παρουσιάσεις και ανταλλαγές απόψεων επί τριών εκθέσεων. Προτείνω καταρχάς να ξεκινήσουμε το σημείο 4, έκθεση Αλφόνση, όσον αφορά τη συμφωνία συνεργασίας, ε, όσον αφορά την Αλία με το Μαρόκο. Κύριε Σιγητά, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αυτή η αλληλευτική συμφωνία με το Μαρόκο αφορά Μία από τις βασικές συμφωνίες που συνήψε η Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα και είμαστε σε μια διαδικασία εγκρίσεως, δηλαδή συνήφθη η συμφωνία και ζητήθηκε η έγκριση αυτής. Αντίθετα με την προηγούμενη φορά που ήταν δευτερευούς σημασία οι συμφωνίε στον αφορά τον όγκο και δεν δημιουργούνταν σημαντικά πολιτικά προβλήματα. Πιστεύω ότι η έκθεση για το Μαρόκο δημιουργεί προβλήματα όγκου και πολιτικά προβλήματα, δημιουργεί πολιτικό πρόβλημα σημαντικό. Δηλαδή ξεπέρασμα του προβλήματος της Δυτικής Σαχάρας μέσω αυτών των σχέσεων ε, και ξέρουμε τι προβλήματα υπάρχουν σε αυτή τη ε, ζώνη και τι γίνεται τον ΟΗΕ. Και είναι πολύ ενοχλητικό αυτό διότι θεωρούμε ότι είναι αντίθετο να, να παραβιάζουμε το διεθνές δίκαιο. Αντιστοιχεί σε αυτό. Δεύτερο, 25% των πιστώσεων αφορά αυτή τη συμφωνία όσον αφορά την πολιτική συνεργασία και εμπορίου και 25% των πιστώσεων είναι πολύ ψηλό και εδώ και αρκετούς μήνες τελούμε αναμονή προβληματισμού επί της ουσίας για την έκθεση, δηλαδή πώς να βελτιώσουν το περιεχόμενο για το περιβάλλον, Όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα επίση πώς να βελτιώσουμε το περιεχόμενο, όσον αφορά την υποστήριξη ανάπτυξη των πλέον ε, των περιοχών που βρίσκονται στην πιο δυσχερή θέση. Λοιπόν, στα συμπεράσματα καλείται η Επιτροπή Αλία να προτείνει στο Κοινοβούλιο την απόρριψη του πρωτοκόλου και μετά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κληθεί να ετοιμάσει ένα νέο πρωτόκολλο λαμβάνοντας ε, υπόψη κάποια αντιστάθμιση όσον αφορά το περιβάλλον και οικονομικά, οικονομική αντιστάθμιση για την ανάπτυξη περιοχή και θα πρέπει να είναι σεβαστέ οι διεθνεί υποχρεώσει όσον αφορά τη Δυτική Σαχάρα. Ευχαριστώ. Δεν ζητάει άλλο το λόγο. Η κυρία Ντεορτή θα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όσον αφορά λοιπόν τις διάφορες θέσεις, σε ένα κοινοβούλιο όλες οι θέσεις είναι νόμιμες, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε κάπως αυστηροί όσον αφορά τις δηλώσεις που γίνονται σε ένα νομικό περιεχομένου κειμένου και όσον αφορά τη δυνατότητα λήψης αποφάσεων όπως είναι αυτή που θα πρέπει να λάβει η Επιτροπή Προπολογισμών. Με κάθε σεβασμό προς τον αξιότιμο κύριο Αλφωσή, στην πρόταση νομίζω ότι μειγνύονται τόσα πολλά στοιχεία και πολιτικά κριτήρια, νομικά κριτήρια και τοποθετήσει Επιτροπής Προπολογισμών που αυτό το έγγραφο ε, δημιουργεί μια τελική, τελικά μια σύγχυση και κατά την άποψή μου δεν πετυχαίνουμε τίποτα εκτός από μια πολιτική τοποθέτηση που κατά την άποψή μου δεν είναι σωστή. Εν πρώτης δεν θέλουμε να εγκρίνουμε ε, την παράταση μιας ελευθερικής συμφωνίας. Δεν πρόκειται περί αυτού, δεν πρόκειται περί θέμα ε, το να σταματήσει η απεικιοκρατία ή να λυθούν πολιτικά προβλήματα. Προβλήματα πρέπει να επιληθούν στον ΟΗΕ και το Κοινοβούλιο είναι υπέρ του να σταματήσει η επικιοκρατία στη Δυτική Σαχάρα. Περιτεύει να αναφέρω ότι πρόκειται περί παλαιάς ισπανικής απικίας. Αλλά σήμερα είναι μία αυτόνομος περιοχή που ε, έχει υποστεί ένα καθεστώς απεικιοκρατίας. Λοιπόν, δεν σεβόμαστε το κριτήριο το σωστό. Δηλαδή, ποια κριτήρια πρέπει να γίνονται σεβαστά για την αληθική συμφωνία. Βασιζόμαστε στα ήδη βιστάμενα πρωτόκολλα και πάντα σεβαζο, σεβόμασταν σαν Ευρωπαϊκή Ένωση τη συμφωνία σύμφωνα και με την άποψη των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου. Πάντα προσπαθούσαμε να σεβόμαστε το διεθνέ δίκαιο. Το μόνο απαιτεί το διεθνέ δίκαιο για να μην αποτελεί απικία μια περιοχή και να σεβόμαστε και το δικαιώματα του πληθυσμού είναι η συμφωνία να ωφελεί τον πληθυσμό και την περιοχή Μέχρι τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδινε χέγγια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με τα οποία η περιοχή αυτή θα έλεγα περισσότερο η χώρα που δικεί αυτή την περιοχή με νόμιμο τρόπο ή μη νόμιμο τρόπο αλλά που δικεί de facto αυτή την περιοχή, αυτή η χώρα ε, να κινείται με τρόπο που να ωφελεί και τον πληθυσμό της Δυτικής Σαχάρας. Αυτές είναι οι πληροφορίες που μας έχει δώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει να την εμπιστευτούμε όσον αφορά την απόφαση θα πάρουμε στην Επιτροπή Προπολογισμών. Για το δίκαιο, αν παραβιάζεται το διεθνές δίκαιο είτε ή όχι, δεν μας αφορά εμάς. Υπάρχει το Συμβούλιο της εταιρική Σχέσης που ελέγχει τις διάφορες νομικές πτυχές. Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ζητά αυτά τα κέρδη, τα ωφέλη να είναι κέρδος του, του ντόπιου πληθυσμού. Δεν είναι σωστό αυτό που αναφέρεται στην έκθεση ότι παραβιάζεται το διεθνές δίκαιο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν συζητούμε να σταματήσει η πιοκρατία η κατοχή αν θέλετε της Δυτικής Σαχάρα, Μιλάμε για μια αληφτική συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεω και Μαρόκου. Και θέλουμε να υποστηρίξουμε και τον πληθυσμό της Δυτικής Σαχάρα μέσα στο σωστό πλαίσιο, στο πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Μετά ο κύριος Αλφωσή, Κύριε Αλφωσή, μάλλον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αξιολογήσει το κόστος αυτής της συμφωνίας αλληλευτικής. 219 άδειε και 25% ή 10% το κόστος δεν είναι σημαντικό. Αυτό είναι κάτι που απορρέα από την διαπραγμάτευση της αλληλευτικής συμφωνίας. Μετά, όταν ζητείτε να υπάρχει κοινή συνεδρία σε Επιτροπής Ανάπτυξης, Επιτροπής Αλίας, για να διαπιστωθεί κατά πόσο προστατεύεται το περιβάλλον και κατά πόσο λαμβάνονται υπόψη οικονομικές πτυχές, και κατά πόσο ωφελείται ο ντόπιο πληθυσμό. Αυτό είναι κάτι που είναι εκτός της, ε, του πεδίου εφαρμογή τη αρμοδιότητα τη Επιτροπή Προπολογισμών. Η Επιτροπή Προπολογισμών πρέπει να εξολογήσει τα περιβαλλοντικά κριτήρια ή θα καθορίσει αυτά που αποφασίζονται στο Συμβούλιο Σύνδεσης όσον αφορά το Εθνές Δίκαιο. Εγώ νομίζω ότι εδώ γίνεται προσπάθεια να χρησιμοποιηθεί το κείμενο για πολιτικούς σκοπούς. Με στρεβλό τρόπο. Δηλαδή η παράταση μιας ε, αλευτικής συμφωνίας χρησιμοποιηθεί για πολιτικούς σκοπούς. Είναι ένα πρωτόκολλο μάλλον θα έλεγα που ζητά την παράταση διαπραγμάτευση μιας αλευτικής συμφωνίας μέσα στην οποία εντάσσονται τα διάφορα εχέγγυα που απαιτούνται ούτω ώστε πραγματικά να γίνεται σεβαστό το διεθνές δίκαιο. Στην Ολομέλεια την πρόσφατη ψηφίσαμε κάτι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την Αλληλευτική Συμφωνία. Συζητήθηκε αυτή η συμφωνία και σε διάφορε επιτροπέ του Κοινοβουλίου. Τοποθετήθηκε η Ολομέλεια. Τώρα καθυστερούμε την έγκριση μιας προσπάθειας που έχει δρομολογηθεί. Θα πρέπει να υπάρξει μια συμφωνία που θα τηρεί καλύτερου, θα περιέχει καλύτερου όρου από την ισχύουσα. Ευχαριστώ κυρία μου, ο κύριος Άγγλουντ έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να πω μερικά λόγια εφόσον είμαι εισηγητή στην Αλληλευτική Συμφωνία, στην Επιτροπή Αλίας για το θέμα αυτό. Οι δύο πρώτες παρεμβάσεις έδειξαν ότι δεν είναι πολύ ευχάριστο καθήκον να είναι κανείς εισηγητής αυτού του χαρτοφυλακίου διότι υπάρχουν πολλά ανάμεικτα συναισθήματα και νομίζω ότι οι συνάδελφοι αυτό έδειξαν πάρα πολύ καλά, ότι αυτό ισχύει. Συμφωνώ με αυτό που είπε ο σοσιαλίστης συνάδελφος όσον αφορά την προσέγγιση, θα πρέπει να κάνουμε εμείς στην Επιτροπή ε, προπολογισμών. Υπάρχουν πολλά περιβαλλοντικά, οικολογικά προβλήματα που περιέχονται στην έκθεση. Δείτε την έκθεση αξιολογήσεως Ε, δείχνει ότι υπάρχουν περιβαλλοντικά προβλήματα, αλλά αυτό δεν είναι βασικό θέμα που απασχολεί αυτή την Επιτροπή. Ούτε θεωρώ ότι είναι βασικό μας καθήκον να αξιολογούμε κατά πόσο η συμφωνία συνάδει με το διεθνές δίκαιο. Δεν είναι αρμοδιότητα της Επιτροπής Προπολογισμών κάτι τέτοιο. Συμφωνώ σε κάποιο βαθμό με αυτό που υπόθηκε για τη Δυτική Σαχάρα, αλλά ήδη η Ολομέλεια με την ε, ψηφο της ε, πλειοψηφίας τοποθετήθηκε. Αλλά βασικό μας καθήκον είναι να αξιολογήσουμε τη συμφωνία αυτή ως οικονομική συμφωνία, διότι είμαστε Επιτροπή Προϋπολογισμών και να δούμε πώς χρησιμοποιούν τα χρήματα του φορολογωμένου. Να παραθέσω κάποια πράγματα από την έκθεση αξιολόγησης της συμφωνίας. Γενικό συμπέρασμα λοιπόν της έκθεσης αξιολόγησης που πρέπει να ετοιμάσει η Επιτροπή για τη συμφωνία ποιο είναι, ότι τα αποτελέσματα τη τετραετία τη αλληλευτική συμφωνία με το Μαρόκο είναι αρκετά απογοητευτικά τα αποτελέσματα τη πρώτη τετραετία. Αυτά ήταν και τα συμπεράσματα χθε που ακούστηκαν όταν συζήτησε η Επιτροπή μα το θέμα αυτό. Δηλαδή, όταν συζητήθηκε το θέμα στην, αλληλευτική, στην Επιτροπή Αλία. Υπάρχουν διαφορετικέ προσεγγίσεις για το πώ να αντιμετωπιστεί το θέμα, όπω ανέφερε η συνάδελφο. Κάποιοι το βλέπουν αυτό σε μεταβατική περίοδο καθοδόν προ καλύτερη συμφωνία, Κάποιοι θέλουν να σταματήσει αυτή η συμφωνία αμέσω, αλλά χτε στην Επιτροπή Αλληλεία εκφράστηκε η άποψη ότι είναι κακή αυτή η συμφωνία και πρέπει να υπάρχει καλύτερη συμφωνία στο μέλλον. Αυτή ήταν γενικά η συμφωνία όλων των συναδέλφων, όλων των πολιτικών ομάδων. Τώρα πώ θα αντιμετωπιστεί το θέμα είναι κάτι διαφορετικό και θα δούμε πώ θα ψηφίσουμε στο τέλο. Θα ήθελα να πω όσον αφορά τα οικονομικά ζητήματα ότι η αξιολόγηση της συμφωνίας από μια οικονομική σκοπιά καταλήγει στο συμπέρασμα ότι από όλες τις συμφωνίες που ισχύουν στην, ε, της Ευρωπαϊκής Ενώσεως εδώ το μεγαλύτερο βάρος τίθεται σχετικά στους Ευρωπαίους φορολογουμένους. Είναι αντικειμενική η έκθεση αξιολόγησης πάνω σε αυτό. Εγώ σας λέω τι λέει η έκθεση αξιολόγησης. Και λέει ότι όσον αφορά το κόστος όφελος στη συμφωνία μεταξύ Μαρόκου και Ευρωπαϊκής Ενώσεως είναι η λιγότερη επιτυχής από όλες τις διμερείς, διμερείς αλληλευτικές ε, συμφωνίες. Αυτά φίλοι μου πιστεύω ότι πρέπει να συζητήσουμε στην Επιτροπή μας διότι αυτό είναι το βασικό μας καθήκον και ελπίζω να προσπαθήσουμε να μην μπούμε στο θέμα αυτό της Δυτικής Σαχάρας. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό θέμα, αλλά όπως γνωρίζουμε δεν μπορούμε να το λύσουμε σε αυτή την Επιτροπή και δεν θα λύσουμε ούτε τα οικολογικά προβλήματα που είναι πολύ δύσκολα ε, με το θέμα των αλληλευτικών αποθεμάτων που ανησυχεί την Επιτροπή Αλίας. Αυτό με ανησυχεί και γι' αυτό θεωρώ, Πρόεδρε, ότι θα πρέπει να τοποθετηθούμε σαφώ επί του θέματο. Είναι μια συμφωνία που οικονομικά δεν είναι βιώσιμη. Αυτό είναι το συμπέρασμα τη έκθεση αξιολόγηση. Και δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε άλλο συμπέρασμα. Για πολιτικού λόγου μπορεί να προσπαθήσει να πει κανεί ότι είναι ένα κακό μήνυμα προ το Μαρόκο να είμαστε σκληρότεροι. Αλλά να θυμηθούμε ότι το 1999 η συμφωνία τερματίστηκε για παρόμοιους λόγους και ήμασταν επί οκταετία χωρίς συμφωνία και το δράμα δεν ήταν πολύ μεγάλο. Η συνεργασία με το Μαρόκο είναι κάτι σημαντικό, είναι εταίρος μας το Μαρόκο ε, γιατί είναι στη Βόρεια Αφρική, θα έπρεπε να ενταχθεί στην πολιτική ε, γυτνίασης αυτή θα πρέπει να ωφελεί και τις δύο πλευρές η συμφωνία. Εδώ δεν ωφελεί τους Ευρωπαίους φορολογούμενους κάποιους τομείς της Ισπανικής αλίας ωφελεί, αλλά όχι γενικά τον Ευρωπαίο φορολογούμενο. Αυτή είναι η άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λοιπόν, όποιος θέλει να δει την έκθεση αξιολόγησης, με τα χαρά να του τη δώσω να τη δει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πιστεύω ότι ακούγοντας αυτά που είπαν οι προτελήσατες συνάδελφοι ε, θα μπορούσαν ε, να επανελειφθούν και από μένα διότι αρμοδιότητες Επιτροπής Προϋπολογισμών δεν είναι να εισέλθει στην ε, ουσία της συμφωνίας. Η Επιτροπή Αλίας καλείται να κάνει κάποιες αξιολογήσεις συγκεκριμένες. Εξάλλου δεν πιστεύω ότι είναι αρμοδιότητά μας να παρέμβουμε για να αξιολογήσουμε το κατά πόσο νομικά είναι συμβατή η συμφωνία όσον αφορά το διεθνές δίκαιο. Και διότι όσον αφορά αυτά τα ζητήματα θεωρώ ότι ήδη υπήρξαν κάποιες νομικές τοποθετήσεις. Το νομικό συμβούλιο του ΙΕ τοποθετήθηκε, η νομική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τοποθετήθηκε. Έχουμε νομική άποψη του Συμβουλίου και έχουμε άποψη και της νομικής υπηρεσίας του Κοινοβουλίου. Δεν νομίζω ότι τώρα η δική μας Επιτροπή θα πρέπει να παρέμβει επ' αυτού και διότι δεν είναι σίγουρα δική μας ε, αρμοδιότητα. Είναι σαφές λοιπόν ότι όσον αφορά τη θέση του συναδέλφου Αλφόνση υπάρχει κάτι πρέπει να επαναξεταστεί. Πιστεύω ότι όσοι πολιτικές ομάδες μπορούν να συνεργαστούν για να επανεξετάσουν αυτά που έγιναν στο σχέδιο κειμένου. Πέραν αυτού θα πρέπει να θυμηθούμε αυτό που είπε κάποιος πριν, ότι το Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια της τελευταίας ολομελίας απέρριψε το ψήφισμα Νταφ, Αλφόνση κλπ. που ζητούσε τη γνωμοδότηση του ΔΕΚ. Πρέπει να το λάβουμε υπόψη αυτό. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να ξανακολουθήσουμε τη διαδρομή που ήδη έχει γίνει, διότι εξάλλου η παρέμβαση του δικαστηρίου δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι πάρα πολύ χρήσιμη, δεδομένου ότι η παράταση της συμφωνίας θα λήξει 17 ε, Φεβρουαρίου 2012. Κατά την άλλη πλευρά το δικαστήριο σίγουρα σε αυτό το χρονικό διάστημα θα δώσει καμία απάντηση. Δεν νομίζω ότι θα είναι λύση λοιπόν αυτό ότι μπορεί να δώσει μεγαλύτερη σαφήνεια απόφαση του δικαστηρίου. Θα καλέσω τον συνάδελφο Αλφονσή να λάβει υπόψη αυτά που διαφάνησαν από αυτή τη συζήτηση για μια επανεξέταση της γνωμοδοτήσεως που παραμένει και να παραμένει περιορισμένη στην αρμοδιότητα τη Επιτροπή Προπολογισμών και να μην ξεπερνάει τα όρια των αρμοδιοτήτων τη Επιτροπή. Ευχαριστώ. Η Εστέλ Γκρελιέ έχει το λόγο τώρα. Καταρχήν θα πρέπει να μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ποια είναι η δυνατότητα που έχει για χειρισμούς και ποιες θα είναι και οι επιπτώσεις διότι ε, τελικά αντιλαμβανόμαστε ότι επεμβαίνουμε 8 μήνες μετά την έναρξη της συμφωνίας ενώ θα έπρεπε να αναδιαπραγματευτούμε την επόμενη συμφωνία η οποία θα ισχύσει από του επομένου Φεβρουαρίου. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν τις προθεσμίες αυτές και θα ήθελα να μου τις διευκρινίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως είπε ο κύριος Αλφόνση το πρωτόκολλο αυτό είναι, δεν είναι ικανοποιητικό αλλά ε, πρόκειται για μία ε, αλληλεία την οποία προσπαθούμε να αναβαθμίσουμε και ελπίζω ότι θα μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν οι διαδικασίες για την έγκριση για να μην αμφισβητούμε τα πάντα ε, ε, κατόπιν γεγονότος όταν όλα θα έχουν αποφασιστεί. Κύριε Χάγκλουν, θέλετε να απαντήσετε στην κυρία Γκρελιέ, όχι? Εσείς ζητήσετε το λόγο για να απαντήσετε στην κυρία Γκρελιέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Διάφορα σχόλια σχετικά με τον φάκελο αυτό. Δεν συμφωνώ καθόλου με τον κύριο Αλφόντσι. Καταρχήν όσον αφορά τη μορφή και νομίζω ότι εδώ η διατύπωση δεν είναι σαφής διότι μετά από το σκεπτικό στην τρίτη παράγραφο βλέπουμε ουσιαστικά ότι ξεκινούμε με τις ε, επιπτώσεις. Άρα ε, εδώ η ουσία δεν μας βρίσκει σύμφωνος. Είμαστε δημοσιονομική αρχή και δεν υπάρχει κανένα δημοσιονομικό επιχείρημα για να καταψηφίσουμε ε, τη συμφωνία αυτή με το Μαρόκο. Ε, το μόνο το οποίο λέγεται είναι ότι θα μας προσφέρει 36,1 εκατομμύρια ευρώ. Μόνο αυτό. Τα άλλα δεν ξέρουμε και ότι θα αντιπροσωπεύσει 25% του σχετικού κονδυλίου του προπολογισμού είναι μια σημαντική συμφωνία που έχει διάφορα συστατικά στοιχεία τα οποία επηρεάζουν και το κονδύλι του προπολογισμού δεν είναι τόσο μεγάλο ε, κατά τρόπον ώστε να ε, απορρίψουμε αυτή τη μεταφορά. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω αν υπάρχουν άλλες ε, δημοσιο νομικές ε, αιτίες για την οποία θα απορρίψουμε αυτή τη μεταφορά. Δεν συμφωνώ λοιπόν. Δεν νομίζω ότι πρέπει να αντιταχθούμε σε αυτή τη ε, μεταφορά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκαρίγκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τα επιχειρήματα ήδη εκτέθησαν και δεν ε, χρειάζεται να κάνουμε ισπανική συζήτηση και εγώ συμμερίζομαι τα επιχειρήματα ορισμένων συναδέλφων και ίσως να μην έχει και πολύ νόημα να συνδέουμε ορισμένες πτυχές όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα με την αλληλεία. Πιστεύω ότι ως Επιτροπή Προπολογισμού ανέκαθεν είχαμε εισηγητές για την αλληλεία που δεν συνέχεια τα θέματα αυτά. Νομίζω πως το καλύτερο θα ήταν να μην ακολουθήσουμε αυτή τη σύσταση και να ψηφίσουμε μάλλον και να απορρίψουμε αυτήν τη σύσταση αντίθεσης προς την Συμφωνία Αλίας και για τους λόγους που εξέθεσαν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Μάλιστα, κύριε Άγκλουντ, θέλετε να πάρετε το λόγο και βεβαίως ο κύριος ηγητής θα ολοκληρώσει στη συνέχεια. Ο κύριο Άκλοντ, καταρχήν, η κυρία Γκριλιέ βγήκε, αλλά ήθελα να πω ότι ο αντίκτυπο θα είναι πως θα πληρώσουμε για το χρόνο που περάσαμε φέτος η παράταση είναι για ένα χρόνο, δηλαδή μέχρι το Φεβρουάριο, δηλαδή μέχρι ότου ψηφίσουμε στην Ολομέλεια που πιθανότατα θα γίνει τον ε, Ιούνιο, γιατί οι διαπραγματεύσεις για ένα κοινό ψήφισμα σε μια, στην Επιτροπή Αλλιές ήταν ιδιαίτερα επικριτικές και υποδείξαμε ότι πρέπει να αλλάξουμε πράγματα στη συμφωνία. Άρα λοιπόν θα ψηφίσουμε τον ε, Ιανουάριο, άρα μόλις ένα μήνα πριν από το τέλος της περίοδου, έτσι κι αλλιώς. Αυτό σημαίνει ότι αν ψηφίσουμε όχι και έπειτα πληρώσουμε για 11 μήνες αντί για 12 μήνες δεν έχει και μεγάλο νόημα. Ούτως ή άλλως θα πληρώσουμε. Στην πράξη δηλαδή αυτό είναι το μόνο, η μόνη αλλαγή. Οι οικονομικές πτυχές πραγματικά πολύ θα ήθελα να είχατε ακούσει αυτά που είπα πριν για την ε, ε, έκθεση αξιολόγηση για τι οικονομικέ πτυχέ. Αυτό πρέπει να το συζητήσουμε. Αν απλώ ψηφίσουμε ναι, σημαίνει ότι θα έχουμε έκθεση αξιολόγηση. Η Κομισιόν πρέπει να την κάνει. Ε, καταλήγει στο ότι δεν είναι βιώσιμη από οικονομική άποψη αυτή η συμφωνία. αν το δεχτούμε θα σημαίνει ότι δεχόμαστε εμεί η Επιτροπή Προπολογισμού τη κακή δαπάνη ε, των δημοσίων χρημάτων και θα σα τα στείλω σε όλου την αξιολόγηση αυτή. Και δεν είναι δικέ μου απόψει. προέρχονται από μια αντικειμενική έκθεση αξιολόγηση την οποία μπορείτε να μελετήσετε όλοι σας. Αυτή είναι η οικονομική πτυχή και φυσικά θα υποβάλω τροπολογίες για να μπουν όλα αυτά στην έκθεση, γιατί νομίζω αυτή είναι η δουλειά μας, να δούμε, να εξετάζουμε τις οικονομικές πτυχές της ε, συμφωνίας. Και αυτές είναι πολύ προβληματικές. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Κύριε Σιγητά, και εσείς ποια πορίσματα φτάνετε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να σας πω ότι δεν είναι ούτε δικό μου ούτε δικό σας λάθος εάν ε, επιλαμβανόμαστε μία συμφωνία η οποία έχει γίνει εδώ και πολλούς μήνες και ε, θα εκπνέει όταν ε, θα ψηφίσει το Κοινοβούλιο αλλά σύμφωνα με το σκεπτικό αυτών οι οποίοι ε, έθεσαν το πρόβλημα θα πρέπει να αποδεχόμαστε τα πάντα να αφήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει ό,τι θέλει και εμείς απλώς να επικυρώνουμε. Δεν συμφωνώ όμως ότι αυτή είναι η σωστή οδός. Πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας γιατί η έκθεση αυτή είναι σημαντική και η Επιτροπή μας είναι υποχρεωμένη να το εξετάσει και αυτό την υποχρεώνεται μάλιστα από τις αρχές οι οποίες ε, επεμβαίνουν για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τους οικονομικούς πόρους ε, προσεκτικά και ε, να εξετάσουμε την τακτικότητα των δαπανών. Εδώ μας ζητείτε να κάνουμε δαπανών δαπάνες, πράγμα το οποίο μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα ακόμη και στην Επιτροπή Υπολογισμού. Δεν αναφερόμαστε μόνο στην τακτικότητα των δαπανών, αλλά και το στόχο. Ο στόχος της βιώσιμης ανάπτυξης είναι κάτι το οποίο πρέπει να επαληθεύουμε. Πρέπει να δούμε αν αυτό εκπληρώνεται με τις αποφάσεις που μας ζητείτε να αποδεχθούμε. Ε, θα ήθελα ίσως να έρθει ο υπεύθυνο αλίας να μας εξηγήσει την ουσία του προβλήματος διότι βλέπουμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα και το κατά πόσον συνάδει με την βιώσιμη ανάπτυξη την οποία έχουμε σχεδόν ομόφωνα υπερψηφίσει. Θα ήθελα λοιπόν να ευχηθήσω την προσοχή όλων των συναδέλφων στην ε, ε, συμφωνία αυτή. Ε, το να αφήσουμε απλώς να προχωρήσουν τα θέματα στην νότια όχθη της Μεσογείου είδαμε που μας οδήγησε στην την Ισία, στη Λιβύη και σε άλλες χώρες οπότε εάν απαρνηθούμε τις αρχές μας κάνουμε έναν πολύ κακό υπολογισμό για το μέρον και για για περιβαλλοντολογικούς και πολιτικούς λόγους ε, λυπάμαι αλλά ε, και ε, το δημοσιονομικό σκέλος είναι πολιτικό σκεπτικό και πιστεύω ότι πρέπει να υπενθυμίσει το κοινοβούλιο στις στα άλλα θεσμικά όργανα ότι πρέπει να σέβονται τη δημοκρατία. Ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή η, με η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων δεν έχει αναλάβει να διατυπώσει μία γνωμοδότηση, κύριε Χάγκλουντ, όχι. Και, κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Χάγκλουντ. Νομίζω ότι θα ήταν σκόπιμο αυτή τη στιγμή διότι εδώ υπάρχουν δύο απόψεις και πιστεύω ότι ε, η η ε, πλειοψηφία στην ψηφοφορία στο περασμένο Στρασβούργο απέδειξε ότι δεν υπάρχει νομικό πρόβλημα και ε, δεν ζητήθηκε η γνωμοδότηση της ε, ε, Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων που θα ήταν χρήσιμο. Υπάρχει το θέμα της Δυτικής Σαχάρας. Ξέρω ότι ο εισηγητής αγαπά πολύ το θέμα αυτό αλλά δεν μας οδηγεί προς ένα. Έχουμε μία γνωμοδότηση από την Επιτροπή Ανάπτυξης, από τη δικιά μας Επιτροπή και ε, μετά στην επανεξιολόγηση θα υπάρξει μία γνωμοδότηση για τις εξωτερικών υποθέσεων αλλά θα είναι πολύ αργά. Ευχαριστώ τους εισηγητές και νομίζω ότι η κατάληξη στην οποία να πρέπει να οδηγηθούμε είναι ότι κάθε φορά που υπάρχει μία ενέργεια σε ένα χώρο εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως καλό είναι να έχουμε την έμπειρη γνώμη της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων ε, διότι η πολιτική είναι η ουσία αλλά εμείς δεν είμαστε ειδικοί των εξωτερικών υποθέσεων υπάρχει μια κατάλληλη επιτροπή, μια αρμόδια επιτροπή και αυτό είχε γίνει με το πρόβλημα της Παλαιστίνης προτού ε, λάβουμε θέση εργαστήκαμε στενά με την ε, Επιτροπή Αναπτύξεως και μάλιστα από κοινού ε, επισκεφθήκαμε τη χώρα για να δούμε πώς προχωρούν οι Ισραηλοπαλαιστινιακές διαπραγματεύσεις να το ίδιο θα έπρεπε να γίνει και με την κατάσταση της Σαχάρας και πόσο επηρεάζει αυτό την ε, συνθήκη αλληλείας και καλό θα ήταν να έχουμε την έμπειρη γνώμη της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, πράγμα που θα θίξω στην επόμενη συνεδρίαση των ε, Προέδρων των Επιτροπών. Ε, έχουμε ε, την την ψηφοφορία για το θέμα αυτό το Νοέμβριο και τώρα θέλω να δώσω το λόγο εις ε, τον ε, Γκόραν Βέ για την αίτηση της Κροατίας να γίνει μέρος Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ναι κύριε Πρόεδρε, ξέρετε ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία η οποία πρέπει να κυρωθεί τώρα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από τις ε, ε, από τα κράτη-μέλη και θα γίνουν δύο εκθέσεις, ένα επίσημο και ένα κατά πρωτοβουλία για τα, τις πολιτικές επιπτώσεις και εμείς πρέπει να γνωμοδοτήσουμε για αυτή τη δεύτερη έκθεση. Η ιδέα είναι ότι θα πρέπει να ψηφίσουμε την έκθεση αυτή κατά τρόπον ώστε ώστε να μπορέσει να ψηφιστεί ε, στην Ολομέλεια το Νοέμβριο διότι υπάρχουν αρχές Δεκεμβρίου εκλογές στην Κροατία άρα θα μπορέσουν να λάβουν μία απόφαση με τη νέα κυβέρνηση πριν τα Χριστούγεννα και μέχρι το, την 1η Ιουλίου 2013 να μπορέσουν να προσχωρήσουν. Ε, βασιζόμαστε εδώ τα απορίσματα της αντιπροσωπείας της κοινή Επιτροπής ε, μεταξύ δύο επιτροπών οι οποίες δεν είχαν μεν συμφωνήσει πλήρως αλλά νομίζω ότι σε γενικές γραμμές ε, ε, συμπλέαμε εδώ ασχολούμαστε μόνο με οικονομικά ε, και δημοσιονομικά θέματα. Υπάρχουν ορισμένα σημεία που δεν συμφωνούμε, όπου η Κροατία πρέπει να επιμείνει, αλλά όχι στο βαθμό ο οποίος πρόκειται να διακυβεύσει την ε, συνέμεσή μας στο να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμη όμως ε, και αν την αποδεχτούμε... δεν σημαίνει ότι όλα βαίνουν καλό στην, ε, στην Κροατία. Στο σημείο 3 λέμε ότι χρειάζεται εξυγχρονισμός της οικονομίας, περαιτέρω, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και διαφοροποίηση. Διότι αυτό είναι το πρόβλημά τους. Εξαρτώνται αποκλειστικά και μόνο από τον τουρισμό. Πρέπει να διαφοροποιήσουν την οικονομία τους, να, ε, χρησιμο... Ε, να προβλέψουν χρήση διαρθρωτικών ταμείων για να επιτύχουν αυτή τη διαφοροποίηση. Τέλος, ε, ε, αυτό ήταν ένα από τα απορίσματα της αντιπροσωπείας. Ανησυχούν για τη δυνατότητα ε, αφομοιώσεως της Κροατίας και τις διαχειριστικές δυνατότητες, διότι εδώ θα μιλάμε μετά την προσχώρηση για πολύ μεγαλύτερα κεφάλαια. Πρέπει λοιπόν πέραν της κυβερνήσεως να αναπτυχθούν Λοιπόν, σε περιφερειακό και σε τοπικό επίπεδο ο δυνατότητες αφομοίωσης οι οποίες προς το παρόν είναι περιορισμένες. Πέραν αυτού θα πρέπει να στηρίξουμε τη δημιουργία μιας προσωρινής οικονομικής βοηθείας και του σχετικού μηχανισμού κατά τρόπον ώστε να ενισχυθεί ε, πρώτης προσχωρήσεως η δυνατότητα εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας ή στη διοικητική στο διοικητικό και τον δικαστικό τομέα στην Κροατία να ε, ξαναεξετάσει ε, το ε, σχετικά με την προσωρινή δυνατότητα στο Σέγγεν εάν μπορεί να συντηρήσει και να ενισχύσει τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και κάποια στιγμή να προσχωρήσει στο σύστημα Σέγγεν και τέλος όσον αφορά τη διαφθορά ίσως γνωρίζετε ότι έχουν κινηθεί κατά πολύ, ε, ε, πολύ ισχυρών πολιτικών, πρώην πρωθυπουργών, υπουργών κτλ. με μεγάλη αποτελεσματικότητα. Παραμένει όμως ένα πρόβλημα στον τομέα αυτό στην Κροατία διότι η διαφθορά δεν είναι μόνο στο ύψιστο επίπεδο αλλά σε όλους τους τομείς της ε, κοινωνίας πρέπει να καταπολεμηθεί η διαφθορά και εμείς πρέπει να προστατεύσουμε τα οικονομικά συμφέροντα και τα δημοσιονομικά συμφέρεια και το συζητούσα με τον πρέσβη προ ε, ε, ημερών αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει απόδειξη ε, ούτε μία περιπτώσεως διαφθοράς που να αναφέρεται σε θέματα κυβερνητικών πόρων, ε, ε, κοινοτικών πόρων. Τέλος, ε, οι δημοσιονομικές προοπτικές. Πώς θα αντιμετωπίσουμε την ε, Κροατία μετά το 2007 από όταν ξεκίνησε αυτός ο προπολογισμός δεν είχαμε λάβει υπόψη την προσχώρηση της Κροατίας και το Συμβούλιο των Υπουργών εξέτασε το θέμα και θεώρησε ότι θα πρέπει να υπάρχει μία αναδιάταξη ε, του προϋπολογισμού για να περιλάβει την προσχώρηση της Κροατίας. Είναι όμως εκατοντάδες εκατομμυρίων και εδώ παλεύουμε όταν μιλάμε για δεκάδες εκατομμυρίων το θέμα είναι δύσκολο αν πρέπει να υπάρξει μία αναδιοργάνωση ε, θα ξεπεράσουμε και το 2013 και θα πρέπει να αναμορφώσουμε και την επόμενη δημοσιονομική περίοδο και πέραν ε, των ε, οικονομικών πτυχών ε, είναι δύσκολο να πούμε στην Κροατία πολιτικά ότι δεν έχουμε επαρκή χρηματοδότηση για να χρηματοδοτήσουμε την προσχώρησή σας ιδίως όταν βρίσκονται προ ενός δημοψηφίσματος το οποίο κατά πάσα πιθανότητα θα έχει αίσια έκβαση αλλά όχι με μεγάλη πλειοψηφία. Άρα αυτό που προσπαθούμε να πούμε στις παραγράφους 8 μέχρι 12 είναι ότι χρειάζονται δημοσιονομική δυνατότητα και καλούμε την Κροατία να συμμετάσχει στο ε, επόμενο ε, δημοσιονομικό προγραμματισμό κατά τρόπον ώστε να συμμετάσχουν και στις διαπραγματεύσεις. Αυτή είναι η πρότασή μας. τότε ευχαριστώ κύριε έχουν ζητήσει δύο το λόγο. Η Ίνγκε Κρέσλε. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι η γνωμοδότηση του Γκέρεντ είναι πολύ καλή. Ε, είχα μία ευχάριστη έκπληξη πρέπει να σας πω. Αλλά θα ήθελα να αναφερθώ στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ε, ήδη με μια παλιά χώρα την Ελλάδα στο θέμα της διαφθοράς και της δικαιοσύνης και το βλέπουμε ε, και στις χώρες που είναι νέα μέλη όπως η Βουλγαρία Ρουμανία. Δηλαδή πιστεύω ότι η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν έπρεπε να, είναι, να έχει μια τόσο ρόδινη διατύπωση ε, και καλό θα ήταν να καλέσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, να διατυπώνει εκθέσεις όπου να διαφαίνονται σαφέστερα οι ε, πρόοδοι διότι στην Κροατία υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στην απονομή δικαιοσύνης και εκπλησώ διαρωτώμεθα πάντοτε Άρα ελπίζω ότι κάθε φορά που έχουμε μία έκθεση για την ε, καθυστέρηση θα είχαμε και μία αναφορά του τι διορθώθηκε εντωμεταξύ για να υπάρχει μία θετική πίεση η οποία θα εξασκείται. Και θα ήθελα να προσθέσουμε μία φράση σχετικά με την βελτίωση της ενημέρωσης ως προς τις προόδους για να ξεχωρίζουμε πότε υπάρχει υπάρχει πρόοδος και πότε οπισθοδρόμηση, το οποίο είναι σημαντικό για να ε, διεξάγουμε μία ύψιστη εξωτερική πολιτική. Ευχαριστώ. Όπως βάζουμε σε δοκιμές αντοχής στις τράπεζες θα πρέπει να υποβάλουμε και τις χώρες σε stress test όσον αφορά την τιμιότητα και τη διαφορά. Ε. Αλλά με κριτήρια πιο σοβαρά από τα stress test ε, των τραπεζών. Η κυρία Γένσκι. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Φέρο. Ε, έξοχη η παρέμβασή του σαν φατοσχέδιο Λίγο χρόνο είχα δυστυχώς για να δω ποιες είναι οι δημοσιονομικέ συνέπειε της προσχωρήσεω της εντάξεω τη Κροατία. Μερικά σχόλια έχω. Πρώτον, προσωπικά. Ελπίζω η Κροατία να δημιουργήσει διοικητικές δομές που θα είναι λειτουργικές για τη διαχείριση και τον έλεγχο των ευρωπαϊκών πόρων. Εδώ υποστηρίζω την πρόταση της κυρίας Γκρέσλε πλήρω. Δεν πιστεύω ότι χρειάζεται σειρά κινήτρων και ποινών γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να χρησιμοποιείται υπερβολικά και αυτό είναι παρακινδυνευμένο. Όμως παρόλα αυτά πιστεύω ότι βατικά μέτρα ίσως τελικά να έχουν θετικές επιπτώσεις. Ανησυχώ μήπως η ένταξη της Κροατίας στο τελευταίο εξάμεινο του παρόντος δημοσιονομικού πλαισίου δεν λήφθη υπόψη εγκαίρως. Δεν θα πρέπει να χρηματοδοτήσουμε μέσω αναδιπλώσεως των πόρων την ένταξη της Κροατίας. Τη χρειάζεται πάρα πολλά χρήματα. Συμφωνώ ε, με τον εισηγητή. Αυτά είναι τα πρώτα που έχω να πω. Αργότερα όταν θα μπω σε μεγαλύτερο βάθος την έκθεση θα πω περισσότερα. Ευχαριστώ Ναντέζδα, ο κ. Μπόκρος. Ευχαριστώ πολύ, πολύ σύντομα. Υποστηρίζουμε ένθερμα την ένταξη της κουρατίας. Παρόλο που αληθεύει ότι αυτά που συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση του Γιώραν αληθεύουν. Είναι ένα μόνο βήμα η ένταξη της, ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ένα μακρύ δρόμο. Ισχύει και για άλλε χώρε. Υπάρχει διαφθορά και υπάρχει πρόβλημα με το κράτο ε, δικαίου. και περισσότερα προβλήματα εμφανίζονται τώρα που μιλάμε, άρα θα πρέπει να τονιστεί αν όχι υπερβολικά. Είναι ευαίσθητη η ισορροπία που θα πρέπει να εξευρεθεί και είμαι σίγουρο ότι ο Γιώραν μπορεί να το διατυπώσει διόντω. Θα στείλει έτσι το κατάλληλο μήνυμα να μην κάνει να εφησυχάσουν όμω οι χώρες που είναι ήδη μέλη τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Έχω διαφορετική άποψη για το θέμα του προπολογισμού. Συμφωνώ μεν ότι είναι μεγάλο το ποσό. Δίκιο έχει εκεί ο Γιώραν. Δεν θα πρέπει να είναι νέα χρήματα δε στο σύνολό τους. Εν μέρη μπορεί να είναι νέοι πόροι και εν μέρη αναδίπλωση πόρων. Να το έχουμε υπόψη. Δεν βγαίνει απαραίτητα αρνητικό μήνυμα το κάνουμε αυτό. Ξέρουν οι Κροάτες πολύ καλά ότι αυτό συνέβαινε στους δύο τελευταίους γύρους α, ε, ε, εντάξεων. Δεν πρέπει να θεωρηθεί απαραίτητο ότι είναι ένα άσχημο μήνυμα που στέλνουμε. Δεν φαίνεται να επηρεάζει το δημοψήφισμα που θα λάβει η χώρα Δυστυχώς η κρίση στην Ευρωζώνη έχει περισσότερες, ε, αρνητικέ αρνητικές ε, επιπτώσεις στο μυαλό και την καρδιά των κρατών. Διαβάσατε τον κρατικό τύπο, θα δείτε ότι η μεγάλη πλειοψηφία των διανομένων είναι εναντίον και επηρεάζουν αρκετά αρνητικά το μέτωπο αυτό. Αυτό είναι πιο ανησυχητικό από οποιοδήποτε μήνυμα θα στέλναμε εμείς. Αν θέλετε, να το λάβετε αυτό υπόψη, νομίζω ότι το μήνυμα θα μπορούσε να διατυπωθεί σωστά λογικά. Ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφε. Κύριε Ισηγητά, έχετε την τελευταία λέξη. Θα είμαι συντομότατος. Καταρχάς κυρία Γκρέσλε, συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Καλό θα ήταν να υποβάλει μια σχετική τροπολογία. Έχουμε προθεσμία 27 Οκτωβρίου για υποβολή τροπολογιών. Έχετε δυνατότητα λοιπόν. Δεν νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ μας. Το ίδιο ισχύει για την κυρία Ναΐνσκι και τον κύριο Μπόκρος. Η κατάσταση είναι ευαίσθητη, αυτό είναι σίγουρο. Στην Κροατία ανησυχούν πολύ για την οικονομική κρίση στην Ευρωζώνη και στην Ευρώπη και γι' αυτό θέλω να είμαι πολύ ισορροπημένο στην έκθεση να προσέξω τι θα λέμε. Πρέπει να είμαστε επικριτικοί όταν χρειάζεται, αλλά αν υπερβάλλουμε, αυτό θα μπορούσε να έχει αρνητικές συνέπειες και να επηρεάσει αρνητικά την κατάσταση που στην Κροατία. Διότι ελέγχουν διεξοδικότατα ό,τι λέμε και γράφουμε στο Κοινοβούλιο. Αυτό είναι σίγουρο. Παρακολουθούν καθημερινά ποιο λέει τι, ποιο γράφει τι για την Κροατία και αναφέρονται στον τύπο. Πρέπει να είμαστε λοιπόν πολύ προσεκτικοί και δίκαιοι. Και αυτό προτίθεμαι να κάνω. Ευχαριστώ. Γκόραν. Λοιπόν, να σας υπενθυμίσω, όπως είπε ο Γκόραν, ότι η προθεσμία για υποβολή τροπολογιών είναι 27 Οκτωβρίου, θα θετήσουμε την γνωμοδοτησία μας 7 Νοεμβρίου. Η έκθεση θα θετηθεί από την ΑΦΕΤ στις 14 Νοεμβρίου εν ώψη υιοθέτησης ψηφίσματος στην Ολομέλεια για 1η Δεκεμβρίου. Μας υπενθύμισε ο Γκόραν τα διαδοχικά στάδια. Ένταξη, υπογραφή υπογραφή και ένταξη. Είναι σχεδιασμένα για την ώρα αυτά τα βήματα για την ένταξη των φίλων μας των Κροατών. Τελευταίο σημείο. Ξαναρχόμαστε στη Μπάρμπαρα, η οποία είναι πολύ απασχολημένη με τον ε, συντονιστή της, η οποία θα μας παρουσιάσει δύο σχέδια για κινητοποίηση του Ταμείου για την Παγκοσμιοποίηση ένα για την Αυστρία και ένα για την Ελλάδα. Κυρία Εισηγήτρια, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομη. Χαίρομαι που βλέπω πόσο πίσω από μερικά λεπτά ήταν στο επίκεντρο θερμή σε αυτό το ταμείο και τώρα εξακολουθούμε να θέλουμε να είμαστε κοντά. Ε, τώρα που θέλουμε να είμαστε κοντά στους πολίτες Ευρώπης είναι, δεν είναι κανείς στην αίθουσα. Όλοι που ήταν εναντίον πριν τώρα απουσιάζουν την αίθουσα. Το ΕΡΚ είναι υπέρ της, του Ταμείου, αλλά όσον αφορά την αλληλεγγύη ε, για τους πολίτες υπάρχει η Γιούτα και ο Φάρμ. Είναι οι πυλώνες ε, των σοσιαλιστών σε αυτή την ε, επιτροπή. Σύντομη παρένθεση, διότι απογοητεύτηκα κάπως από την ψηφοφορία που έλαβε χώρα πριν, που ήμασταν όλοι μαζί. Τώρα εδώ μιλάμε για κινητοποίηση πάντα αυτού του ταμείου με πολύ μικρότερα ποσά για δύο χώρες που δεν είναι λιγότερο σημαντικές από τη Γαλλία, διότι το πρώτο αίτημα προέρχεται από την Αυστρία. Οι απολυμμένοι εργαζόμενοι που ζήτησαν τη βοήθεια είναι 502 που ανήκουν σε 706 επιχειρήσεις που λειτουργούν στον τομέα των μεταφορών. Το ποσό είναι 3.640.000 περίπου ευρώ. Δεύτερο αίτημα από την Ελλάδα υποστήριξη 642 εργαζομένων της επιχειρήσεων που είναι στο τομέα του, του λιανικού εμπορίου. Το ποσό είναι 2.900.000 ευρώ περίπου Αυτά είναι, δεν ξέρω αν ε, θέλουν να υποβάλουν τροπολογίες και για τα δύο αυτά αιτήματα συνάδελφοι. Υπενθυμίζω όμως 20 Οκτωβρίου προθεσμία για τις τροπολογίες. 7 Νοεμβρίου θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή Προϋπολογισμών και στην Ολομέλεια τον Νοέμβριο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κύριε Συγήτρια. Ε, υπάρχει κάποιος που θέλει να παρέμβει, να υποβάλει ερωτήσεις στην εισηγήτρια όσον αφορά αυτά τα θέματα. Δεν νομίζω. Λοιπόν, υπενθυμίζω ότι όσον αφορά αυτά τα δύο θέματα έχουν προθεσμία υποβολή τροπολογιών 20 Οκτωβριού η Επιτροπή Απασχόληση θα γνωμοδοτήσει 7 Νοεμβρίου την ίδια μέρα, μερικέ ώρε μετά θα υιοθετήσουμε το σχέδιο έκθεση για να πάει στην Ολομέλεια τον Νοέμβριο. Αγαπητοί συνάδελφοι, Εργαστήκαμε αξιοθαύμαστα την περασμένη εβδομάδα και αυτήν και τελειώνουμε πριν από τις 6.30, οπότε μπορούμε να απελευθερώσουμε ευχαριστώντας τους διερμήνεις και τους συνεργάτες μας και μπορούμε, σας το επιβεβαιώνω, ότι καταργούμε τη συνεδρίαση της Πέμπτης, ακυρώνεται και της επόμενης Δευτέρας. Ε, άρα κάνουμε οικονομίες, δεν κάνουμε δύο συνεδριάσεις, μπορούμε να μπορείτε να ασχοληθείτε με θέματα. Να ευχαριστήσω και τη γραμματεία πριν κλείσουμε, που έκανε δουλειά πάρα πολύ σημαντική, χωρίς την οποία δεν θα μπορούσαμε να κινηθούμε τόσο γρήγορα. Λοιπόν, έληξη συνεδρίαση. Καλό σας βράδυ.